Can I encourage you... Συνάδελφοι, για καθίστε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε κάποτε. Good afternoon, colleagues. Just... Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ξεκινάμε λοιπόν με την αρχή. Υποθέτω ότι δεν έχετε κάποιο θέμα με την ημερησία διάταξη. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις από πλευράς μου σχετικά με τις εργασίες μας αλλά θα πρέπει να τελειώσουμε ακριβώς στις μισή, διότι οι διευμηνείς 6.30 ώρα θα σταματήσουν τις εργασίες. Λοιπόν, έχετε κάποια αντίρρηση για τα πρακτικά. Από το μήνα Φεβρουάριο μέχρι το μήνα Μάιο. Περνάω στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Ε, θα προεδρεύσω κατά τη διάρκεια της εξέτασης του τέταρτου σημείου. Είναι η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας στο ΣΑΕΛ και η συνεισφορά στην ειρήνη και τη σταθερότητα και ασφάλεια του G5 στο ΣΑΕΛ, Μαλή, Μαυριτανία και Νίγηρα. Υπήρξαν επισκέψεις στο Νίγηρα και στο Μάλι το 16 και το 17 διαδοχικά και υπήρξαν αρκετές συζητήσεις για την κατάσταση στην περιοχή και με μέλη των κυβερνήσεων και με βουλευτές και χαίρομαι που έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζακ Φραντά, ο υπεύθυνο για την ολοκληρωμένη στρατηγική προγραμματική πολιτική του EAS. E όπως γνωρίζετε την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Μογκερίνη παρουσίασε την διευκόλυνση την Ευρωπαϊκή για την Ειρήνη. Συνεπώς η συζήτηση την οποία κάνουμε σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σε σχέση με το ερώτημα το οποίο τίθεται, πώς μπορεί δηλαδή το G5, το G5 για το ΣΑΕΛ να υποφεληθεί από την διευκόλυνση αυτή, μιας και έχουμε καθυστερήσει ήδη. Θα σας δώσω κύριε Φραντά αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είμαι μέρος της ε, δομής διαχείρισης κινδύνου και ασχολούμαι με την PSDC. Δεν υπάρχει εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για το γεωγραφικό σκέλος, οπότε δεν πρόκειται ε, να μπω σε ξένα χωράφια. Θα αναφερθώ όμως εξαρτητικά στην κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή του ΣΑΕΛ και τη δράση μας ε, για το ζήτημα αυτό. Ε, Βεβαίω η απουσία των συναδέλφων έχει να κάνει και με το, το γεγονό ότι η κυρία Μογκερίνη σήμερα θα έβλεπε του ε, ε, υπουργού του G5. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποστολή στο Μαλί και στον Ήγηρα, θα σα κάνω μια επικαιροποίηση τη κατάσταση τη ασφάλεια στο ΣΑΕΛ και τη ε, συνεισφορά τη PSDC στην ασφάλεια και την, ε, και την ειρήνη στην περιοχή. Η κατάσταση ό,τι αφορά την ασφάλεια. Ε, θα σα πω τι γίνεται στι διάφορε περιοχέ. Φαίνεται να είναι υποέλεγχο η κατάσταση στο Τσάντ, στο βόρειο Τσάντ και στη Μαυριτανία, όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ασφαλεία. Στον Ήγυρα όμω. Υπάρχει ένα λαθρεμπόριο που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό ζήτημα, υπάρχει ο διάβλος προς τη Λιβύη και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ε, κοντά στη ε, λίμνη την Περίου. Και βεβαίω ε, είναι ακόμα έντονη δράση της οργάνωσης Boko Haram. Ε, πριν από δύο μήνες ε, πρόκειτο να αρθεί η κατάσταση εκτάκτη ανάγκη, τελικά όμως ε, διατηρήθηκε, διατηρήθηκε από την Μπουρκίνα Φάσο μεταξύ των πέντε χωρών του G5 ε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Μπουρκίνα Φάσο είναι η χώρα όπου είναι πιο έστραυστη η κατάσταση από πλευρά ασφαλεία, ιδιαίτερα μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματο, ε, τα συστήματα ασφάλεια και άμυνα τα οποία έχουν πληγεί, αλλά και τι επιθέσει που δέχτηκαν πρόσφατα που ε, καθιστά ακόμα πιο έστραυστη την ασφάλεια. Επίση, το κεντρικό Μαλί ε, κάτι το οποίο βεβαίως πάει και προς τον Ήγηρα και προς την Μπουρκίνα Φάσο, επεκτείνεται αυτή η ανασφάλεια. Γενικά οι παράγοντες ανασφάλεια και αστάθεια ε, ε, κάπως ε, μερικώ μάλλον αντισταθμίζοντα τι προσπάθειε σταθεροποίηση. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Δεν μπορούν να βρεθούν λύσει παρά μόνο σε μια κλίμακα που θα ξεπερνάει την επόμενη γενιά. Χρόνια. Ζητώ συγγνώμη τη Δερμηνή, λέει ο μιλητή. Θα μιλήσω λίγο πιο αργά. Είναι αλήθεια ότι μιλούσε κάπω γρήγορα ο μιλητή. Βεβαίω γαλλικά να μιλήσετε. Κανένα πρόβλημα, αλλά πιο αργά ή δυνατόν. Και συγγνώμη. Θα έρθω τώρα στην περίπτωση του Μαλή. Ε, το Μαλή βεβαίως έχει μια ιδιαίτερη θέση εδώ λόγω του κεντρικού γεωγραφικού του ε, του τοποθέτησης ε, ε, η κατάσταση στο Μαλί δεν είναι και τόσο καλή παρά τις προσπάθειες ε, που έχουν γίνει δεν μπορεί κανείς να είναι ιδιαίτερα αισιοδόξο για το επόμενο έτος στο Μαλί θα λάβουν χώρα προεδρικές εκλογές στις 29 Ιουλίου ενδεχομένως να έχουμε και έναν δεύτερο γύρο 12 Αυγούστου ας δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα εμείς ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και ότι θα έχουμε ένα αξιόπιστο ε, εταίρο μετά από αυτές τις προεδρικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, τρομοκρατικές οργανώσεις που, που ενώνονται ε, εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν τρεις-τέσσερις ε, τρομοκρατικές ομάδες που έχουν συνασπιστεί υπάρχει λοιπόν αυτό ο συνασπισμό των τρομοκρατικών οργανώσεων. Το Μαλή είναι μια χώρα η οποία έχει πληγεί πολύ από την τρομοκρατία και οι δυνάμεις ασφαλείας και άμυνας αλλά και ο πληθυσμό ε, έχουν υποστεί σημαντικέ απώλειε. οι επιθέσεις προς τις στρατιωτικές δυνάμεις ε, πολλαπλασιάζονται και είναι σχεδόν καθημερινέ. Ε, τίνουμε να το ξεχνούμε αυτό έτσι λοιπόν, οι πιο πρόσφατε εξελίξει δείχνουν ότι υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά τι επιθέσει τη Μίνουσρα, η οποία βεβαίω προστατεύεται. Ε, είναι πιο πολύ στο ζητήματα προστασία η συγκεκριμένη δύναμη, ίσω να και ένα χίλιο πτέρνα τη αυτή. Ε, οι επιθέσει κατά του CNS και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ε, ανθρωπιστικών οργανώσεων πολλαπλασιάζονται επίση. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο. 99 επιθέσεις κατά ΜΚΟ και ανθρωπιστικών οργανώσεων το 2017 σε μεγάλη ανωδική πορεία. Οι περισσότερες επιθέσεις συναντώνουν χώρα κυρίως στο κέντρο της χώρας όπου έχουμε και το, το μεγαλύτερο πληθυσμό ε, και βεβαίως είναι και η συνταποθήκη αν θέλετε της χώρας. Η χρηματοδότηση των ομάδων αυτών γίνεται κυρίως από την φορολόγηση διοδίων κατά κάποιο τρόπο, περάσματος, προέρχεται επίσης ε, και από τις απαγωγές ε, δυτικών ε, για τις οποίες ζητούν λίτρα. Τα λίτρα αυτά τους επιτρέπουν να ζήσουν για ένα-δύο χρόνια. Είναι, όπως βλέπετε, μια εξαιρετικά επικερδής δραστηριότητα. Αυτές οι ομάδες μπορούν εύκολα να λαιλατίσουν και να κλέψουν ε, τα περιουσιακά στοιχεία ε, ανθρωπιστικών οργανώσεων, ε, δεν αφήνουν ε, την ανθρωπιστική ενίσχυση να φτάσει στον πληθυσμό, οπότε οι οργανώσει εξαρτώνται ουσιαστικά από τις τρομοκρατικέ ομάδε, είναι αρκετά ανθυγιεινή η όλη διαδικασία. Όλοι ψάχνουν μια νέα, ε, ένα νέο κενό στο δίκτυο ασφαλείας που υπάρχει το βλέπουμε αυτό μετά από αυτό που έγιναν ε, στην πρεσβεία τη Γαλλική στο, στην Μπουρκίνα στο κεντρικό Μαλί οι διεθνικές οι, ε, εντάσεις δεν έχουν εκλείψει με σημαντικές ε, σημαντικά έτσι, βία επεισόδια. Υπάρχουν δημιουργούνται και ομάδες αυτοάμυνας αυτή τη στιγμή επειδή το κράτος δεν μπορεί να υπερασπίσει ε, τους πληθυσμούς, τους, στην, στη Φιλίπ Πέλ, παραδείγματος χάρη, υπάρχει αυτή η, η τάση αυτοάμυνας ακριβώς για να καλυφθεί το κενό που αφήνει πίσω του, το κράτος. Το Μαλί λοιπόν κάνει μεγάλες προσπάθειες, ε, η χώρα, το κράτος του Μαλί προσπαθεί να, να σταθεροποιήσει την περιοχή. Υπάρχει ένα σχέδιο για σταθεροποίηση της περιοχής του κέντρου ε, το οποίο προχωράει σιγά σιγά όμως ε, εξακολουθεί να υπάρχει ένας πυλώνας ασφάλειας πολύ ισχυρός που περισχύει του κοινωνικού πυλώνα και του πυλώνα ενίσχυσης ε, από τον Αύγουστο του 2017 στα πλαίσια μιας δράσης άρθρο 28 δηλαδή χρησιμοποιώντας τον προπολογισμό της ΕΦΣΠ, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για μια δράση σταθεροποίησης στην περιοχή του Μόπτη και Σεγκού για να μπορέσουν να σταθεροποιηθούν οι άλλες τρεις συνιστώσεις αυτού του προγράμματος, δηλαδή διακυβέρνηση, κοινωνικονομική ανάπτυξη και επικοινωνία. Όλες οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας μας έχουν επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε κάπως την κατάσταση, όχι όμως την χώρα. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι ευρωπαϊκές αποστολές, ε, οι ο Κάπ Μαλή, η Μπαρκάν που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο αλλά και διεθνείς δυνάμεις μεταξύ των οποίων η Μιντούσμα ε, ακόμα έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους έως ότι πετύχουν τους στόχους τους έτσι όπως αυτοί έχουν οριστεί. Όπω και να έχουν τα πράγματα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τις τοπικέ πρωτοβουλίες όπω η πρόσφατη πρωτοβουλία διασυνοριακή συνεργασία με βάση το Τσάντ σε σχέση με το ζήτημα της Λιβύης βέβαια δεν είναι κάτι παλαιό. Στις 31 Μαΐου είχαμε μια τριμερή συμφωνία μεταξύ Νίγηρα, Σουδάν, Τσάντ και Λιβύης που υπεγράφει στην Τζαμένα στα πλαίσια της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ε, συνεργάζονται αυτές οι χώρες για να ανταλλάσσουν πληροφορίες, ε, ε, να μπορούν να καταδιώξουν ε, σε μια άλλη χώρα, να υπάρχουν κοινέ περιπολίες και να υπάρχει ένα συντονισμό σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο. Ε, θα είναι κυλιόμενη η διοίκηση, οι δικαστικές αρχές των χωρών που έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία θα πρέπει μέσα σε δύο μήνες να υπογράψουν συμφωνίες ε, δικαστικής συνεργασία για να μπορούν να υπάρχουν και εκδόσει. Ε, στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής έγινε αναφορά και σε προγράμματα ανάπτυξης στις νοριακές περιοχές. Το Τσάντ έχει αναπτύξει περίπου 10 με 15.000 ανθρώπους στην περιοχή του Μπόρκου και του Τσιλαμπέρι. Δεν είναι δηλαδή αμελητές ποσότητες. Τα μεγέθη σε ό,τι αφορά το G5 τώρα πιο συγκεκριμένα, το G5 του Σαέλ, δηλαδή τη περιοχή του Σαέλ και η συνεισφορά του στην ειρήνη και την ασφάλεια. Σε αυτό το δεύτερο κομμάτι θα αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν οι χώρε αυτέ και πώ τη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω σε ό,τι αφορά τη δράση ε, της PSDC, διότι εμείς με αυτό ασχολούμαστε κυρίως. Δεν θέλω να καταστώ έμονος, αλλά θα αναφερθώ στη συνάντηση η οποία έγινε του G5 το Μαλί, το Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρα στο Τσάβ και η Μαυριτανία δημιούργησαν το Φεβρουάριο του 2018 ένα θεσμικό πλαίσιο συντονισμού της περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ανάπτυξης και της ασφάλειας. Ονομάζεται G5 Sahel στο πολιτικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο. Συνδέει την οικονομία και την ασφάλεια και συμμετέχουν όλες οι χώρες του ΣΑΕΛ που ακολουθούν χρηστές μορφές διακυβέρνησης. Η απάντηση βέβαια του ευρύτε, της ευρύτερης ομάδας είναι περιορισμένη διότι δεν υπάρχει ακόμα αρκετή πείρα ιδιαίτερα σε οριζόντιους τομείς στους οποίους υπάρχουν διαφορές πολλές φορές σημαντικότητες. Ο τομέας της ασφάλειας είναι ο μόνος ο οποίος έχει προχωρήσει μέχρι τώρα στα πλαίσια της μικτής δύναμης G5, ΣΑΕΛ, ξεκίνησε στις 2 Ιουλίου του 2017 αυτή η μεικτή δύναμη στρατιωτική ενισχύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης επικυρώθηκε από το ψήφισμα 2359 της, 23ης Ιουνίου του 2017, πρόταση την οποία είχε κάνει η Γαλλία. Η εντολή του G5 Sahel είναι καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού ε, ε, οργανωμένου εγκλήματος και της ε, εμπορίας ανθρώπων. Η πρώτη συνάντηση συνεργασίας έγινε τον Νοέμβριο του 2017. Συμμετείχαν οι πρώτες οι δυνάμεις που προχώρησαν σε αποστολές σε τρεις τομείς γεωγραφικούς, ο πιο δραστήριος είναι ο κεντρικός τομέας, δύο ενέργειες έγιναν στον κεντρικό τομέα και στον ανατολικό τομέα στο Τσάδ και στον δυτικό στη Μαυριτανία προβλέπονται δράσεις για τον Ιούλιο του 18 σχετικά με τις ε, η επιχειρησιακή ικανότητα της δύναμης αυτής θα ολοκληρωθεί ε, σε δύο μήνες. Ε, όλοι κρατούν τις θέσεις τους, δεν αντικαθίσταται η εμισμά των Ηνωμένων Εθνών στο Μαλί, που βοηθούν τις αρχές του Μαλή να σταθεροποιήσουν την χώρα τους. Ε, συνεργάζονται λοιπόν με την δύναμη του ΟΗΕ, η οποία προβλέπει οργανωτική και επιμελητιακή συνδρομή στην δύναμη του G5 Σαέλ. Αυτή η δύναμη των G5 interpretable. Yeah, sorry, it's they are calling that into my ears. Vous avez le temps nécessaire, ne, ne vous inquiétez pas. Oui, je m'excuse encore. Conclusion sur la force G5. Λοιπόν, συμπεράσματα τώρα για την ομάδα των 5. Η μεικτή αυτή δύναμη λοιπόν δημιουργεί πολλές προσδοκίες η πρόταση και για την αστυνομική συνιστόσα. Είναι κάτι για το οποίο πολλά μέλη έχουν αρκετές ελπίδες θα έλεγα, είναι σαφής και τώρα θα πρέπει να γίνει λειτουργική. Ε, σε όλα τα επίπεδα λοιπόν, και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο δικαστικό και σε επίπεδο ποινικό. η λειτουργικοποίηση σε εισαγωγικά της αστυνομικής δύναμης προχωρά με αρκετά υψηλή ταχύτητα και βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως κάποιες δυσκολίες λόγω του νεαρού χαρακτήρα της ομάδας αυτής G5 σε επίπεδο υλικού εξοπλισμού. Ε, λείπει εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακός, επιμελητιακός υποστήριξη των ενόπλων ομάδων, αποθήκευση ε, κτλ. Αυτά λοιπόν απαιτούν εντατικές ε, ε, δράσεις από πλευράς των δωρητριών μεταξύ των οποίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέναντι στις δυσκολίες τις οποίες σας έχω περιγράψει για την λειτουργικοποίηση πάλι σε εισαγωγικά αυτής της ομάδας και της συνιστώσας της αστυνομικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει ανάλογα. Και οικονομική στήριξη και ηλική στήριξη της ομάδας των 5 υπάρχει, προχωρά. Θα υπάρξει επίσης ε, ε, μια ακρόαση στο Σαν Κλού στο Παρίσι που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, για την οργάνωση της στήριξης και μετά από τη συνάντηση η οποία είχε οργανωθεί στις 23 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες ε, με συμπρόεδρους στην Αφρικανική Ένωση, φυσικά την G5 Σαέλ και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη. Θα χρειαστούν περίπου συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία τα 100 εκατομμύρια θα προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Καταπίστευμα για την Αφρική, για την ειρήνευση μάλλον στην Αφρική, για τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων. Όμως η δυσκολία την οποία συναντάμε για να εξοπλίσουμε μια τέτοια δύναμη είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει Αργότερα όταν συζητήσετε για τη συνεισφορά του Νίγηρα στην Διεθνή Δύναμη για την καταπολέμηση του Μπόκο Χάραμ. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα προκαλέσει προβλήματα σε επίπεδο λειτουργία, σε επίπεδο διοικητικό και σε επίπεδο παράδοσης εξοπλισμών. Τώρα, καλύπτουμε λίγο την τον μισθολογικό κενό το οποίο υπάρχει και δίδουμε και κάποια βοήθεια έκτακτη. Έχει ξεκινήσει η συνεργασία αυτή, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Στα πλαίσια λοιπόν του καταλόγου που χρειάζονται για τον σωστό εξοπλισμό του G5, και σε σχέση με τα κράτη-μέλη που θέλουν να πάρουν μέρος ώστε να γίνει η δύναμη αυτή λειτουργική και να διαρκέσει δημιουργήθηκε ένα coordination hub, ένα κέντρο συντονισμού το οποίο λειτουργεί με διάφανο τρόπο και κατανέμει τη βοήθεια σε επίπεδο εξοπλισμών, σε επίπεδο ε, υποδομών και μέσω οδικών ε, τόπων μεταφοράς. Είναι αρκετά περίπλοκο ανάλογα με τα αιτήματα που έχουν αυτοί που ζητούν τη βοήθεια και τις δυνατότητες που έχουν αυτοί που την χορηγούν. Προσπαθούμε να αποφύγουμε κάποιες επικαλύψεις έτσι ώστε να μην χορηγούμε δύο φορές το ίδιο υλικό και θα πρέπει επίσης να αποτρέψουμε και τη διασπορά των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας και να δούμε αν μπορούμε να ενισχύσουμε και την εκπαίδευση. Σε σχέση με το SDC, αυτή τη στιγμή ξεκίνησε υπό την Προεδρία του Μαλή το πρώτο επιχειρησιακό στρατηγείο υπάρχει σωστή συνεργασία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές έτσι ώστε η μεικτή αυτή δύναμη να καταστεί πραγματικά λειτουργική. Σε επίπεδο συμβουλευτικό και κατάρτισης τους βοηθήσαμε ε, να ε, διατυπώσουν ακριβώς ε, τα καταστατικά αν θέλετε έγγραφα να διαμορφώσουν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας της αστυνομικής συνιστώσας Βοηθήσαμε λοιπόν να δημιουργηθεί μια τέτοια δύναμη χωρίς την οποία ε, δεν θα υπήρχαν κάποιες καλές πρακτικές εκ των προτέρων. Αρχικά η δύναμη των πέντε, αυτή η κοινή δύναμη των πέντε ήταν στρατιωτική, αυστηρά, αλλά το Μαλί κυρίως προσπάθησε έτσι ώστε να τεθούν τα θεμέλια μιας ευρύτερης μορφής συνεργασίας. Κάναμε και αρκετά σεμινάρια για την επιμόρφωση των αξιωματικών των αρχηγείων των τριών χωρών, όπως επίσης και για τα στελέχη από πλευρά του Μαλή. Επίσης ενισχύσαμε και την ανακριτική ομάδα της Δημοκρατίας του Μαλή. Ε, εμείς προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε όλες αυτές τις επιμέρους πλευρές. Θέλουμε να υπάρξει σωστός συντονισμός. Αυτή λοιπόν η άμεση προσπάθεια γίνεται ακριβώς μέσω της ενίσχυσης του τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ειδικά στο Μαλί και στο Νίγηρα. Τρεις αποστολές όπως είπα μέχρι τώρα, μία πολιτικής φύσεως εισαγωγικά στο Νίγηρα, μία στρατιωτική και μία πολιτική στο Μαλί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τη Μίνουσμα των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στις τοπικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ κάτι το οποίο θα επιτρέψει στη Μίνουσμα να βοηθήσει σε επίπεδο υποδομών και επιμελητιακό την κοινή ομάδα G5 του Σαχέλ. Και εμείς θα ενισχύσουμε την μήνουσμα συμμετέχοντας στις προσπάθειες ειρήνευσης των πολιτικών δυνάμεων στο Μαλί μετά από τις πρώτες υπογραφές ε, και τα μνημόνια συνεργασίας. Οι προσπάθειες αυτές ε, τίνουν μέσω διμερών τεχνικών συμφωνιών να καλύψουν τα τεχνικά κενά τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά κενά και τέλος, και το είχα πει και πριν 1,5 χρόνο, η περιφερικοποίηση των δράσεων αυτών είναι κάτι το οποίο πρέπει να δείξουμε ε, και στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας πριν από το τέλος του μήνα. Είναι κάτι το οποίο ακριβώς μέσω των αποστολών και δράσεων αυτών να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο και το G5 χωρίς να ξεχάσουμε τη μεικτή δύναμη που ανήκει στο G5 και που είναι ένας από τους στόχους του G5 αλλά δεν είναι αποκλειστικός στόχος. Θα τελειώσω λοιπόν λέγοντας ότι η δράση ασφάλειας και ε, συνεργασίας και άμυνας μάλλον γίνεται σε συνεργασία, σε και με άλλες λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το CSDC και σε συνέργεια με τοπικούς ε, εταίρους όπως Μπαρκάν και τα λοιπά πολλές δράσεις σε επίπεδο λοιπόν του ΣΑΕΛ. Ε, πολλή επιθυμία υπάρχει για συνεργασία και για βοήθεια. και νομίζω ότι όλα αυτά εντάσσονται στην σφαιρική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι δεν σας κούρασα ιδιαίτερα. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και τον κύριο Μπενουά τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε ερωτήσεις από τους συναδελφούς και ελπίζω μετά η Κομισιόν να απαντήσει Βεβαίω και εσεί θα απαντήσετε και κυρίω αυτό μας ενδιαφέρει. Μάικλ, νομίζω εσύ έχεις μια ερώτηση. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Φράντα, για την παρουσίασή σας που μας δίνει μια εικόνα της έθραυστης κατάστασης και τα ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν είναι το που μπορούμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα με τα νέα μέσα που δημιουργούμε όπως η CPSD ή το Αφρικανικό Μέσο για την Ειρήνη. Αλλά πριν έλθω σε αυτά υπάρχει ένα ζήτημα αρχής. η σταθεροποίηση εκεί πέρα επιβάλλεται μόνο από εμάς, την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τη Γαλλία, γιατί το κράτος το ίδιο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, δεν είναι αρκετά οργανωμένο, είναι τόσο χάλια η κατάσταση. Γιατί είχα την εντύπωση πως, ε, δεν ξέρω, οι υπεύθυνοι εκεί δεν μπορούν από μόνοι τους να ανταποκριθούν στον ρόλο τους. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε εμείς ανταυτόν για να υπάρξει κάποια παρουσία κράτους. Επίσης όταν μιλάτε για πολιτικο-στρατιωτική ε, πολιτικο-στρατιωτικό συντονισμό. Ποιος συντονίζει. Και εμείς είμαστε πάλι ή είναι κάποιος από τους πέντε σε θέση να συντονίσει. Δηλαδή, εντάξει, το να το κάνουμε εμείς η Γαλλία συγκεκριμένα βεβαίως με βρίσκει σύμφωνο. Το θέμα λοιπόν είναι τι πρέπει ε, να γίνει έτσι ώστε τελικά να αλλάξει κάτι, να υπάρξει μια σταθεροποίηση τι ε, πρέπει να γίνει, παραδείγματος χάρη, για να σταματήσουν οι παραδόσεις ε, όπλων που μπορεί να καταλήγουν εκεί ακόμα από τα λιβικά αποθέματα ή από τις ακτές. Πώς ε, έχει λοιπόν η κατάσταση. Με τις δυνάμεις που έχουμε και τις δομές που υπάρχουν μπορούμε κάτι να κάνουμε προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάικλ. Και βεβαίως ε, ως πρόεδρος θα κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις μετά τον συνάδελφό μου. Ναι, ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πραντάν για την παρουσίασή του. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και μας επιτρέπει να δούμε ποια είναι πράγματι η κατάσταση στο ΣΑΕΛ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση εδώ, η οποία θα έλεγα με απασχολεί εδώ και καιρό. Εξετάζουμε τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών μονάδων σε αυτό το τμήμα της Αφρικής. Θέλω να θέσω το εξής όμως ερώτημα. Στο συγκεκριμένο αυτό στρατιωτικό πλαίσιο τίθεται κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε το ερώτημα αυτό. Μερικές φορές οι ασκήσεις είναι εύκολες στα γυμνάσια, αλλά φυσικά η πρακτική είναι η δύσκολη. Είναι δυνατόν να εκπαίδευεται κανείς ε, για τις αποστολές αυτές ή μήπως ε, παραμένει το πρόβλημα αυτό συνολικά της εκπαίδευσης για όλες τις ε, δράσεις που αναλαμβάνουμε. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα και συνεχίζοντας την ερώτηση του Μάικλ Είπατε ότι υπάρχουν αρκετές διεθνείς οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται και αναφερθήκατε επίσης στο ότι έχει υπάρξει αρκετός συντονισμός και στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής για την ασφάλεια. Πόσο αποτελεσματικά είναι, οι αποτελεσματικές είναι οι προσπάθειες αυτές. Αναφερθήκατε επίσης και στα θέματα χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων που εκμεταλλεύονται την σώματεμπορία, όπως επίσης και τα έσοδα από απαγωγές. Τι ακριβώς παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή υπάρχουν και σε επίπεδο χρηματοδότησης τις οποίες θα κληθούμε εάν είναι δυνατόν και εμείς να καλύψουμε. Και τέλος στα θέματα χρηματοδότησης είπατε ότι 100 εκατομμύρια από τα υπεσχημένα 400 εκατομμύρια θα προέλθουν από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Σέβονται οι άλλες χώρες τις υποσχέσεις που έχουν δώσει για τα υπόλοιπα 300 εκατομμύρια. Γιατί από ό,τι ακούω υπάρχει μια βραδύτητα για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Έχει υπάρξει κάποια βελτίωση. Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις ε, εξαιρετικά εύστοχες. Υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας. Αν κάνουμε το σωστό και αν κάνουμε τη δουλειά των άλλων επίσης. Ε, εφόσον κατάλαβα καλά το σκεπτικό του ερωτήματος. Από πλευράς CSDP και τα ζητήματα ασφαλείας και άμυνας Όταν ξεκίνησαν οι αποστολές αυτές, υπήρχε ένα δίλημα. Δηλαδή ή έπρεπε να δράσουμε ή να μην δράσουμε. Και αν δεν δράσει κανείς πρέπει να δούμε εκεί ποιο είναι το αποτέλεσμα, ποιες είναι οι επιπτώσεις. Ε, και αν δεν δράσουμε τώρα μήπως είναι πολύ αργά αύριο. Και φτάσαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Ήγηρα μια αποστολή CSDP που ασχολείται ακριβώ με αυτά τα οποία αναφερθήκατε, να βοηθήσουμε δηλαδή τι αρχέ του Νίγηρα ε, στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο. Και όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, βέβαια, ε, εδώ αναφερόμαστε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν ε, ε και του δικού μα συμπολίτε. Ε, λαθρεμπόρια, παράνομη μετανάστευση, τρομοκρατία. Το δίδαγμα λοιπόν είναι ότι Βεβαίω οι τοπικέ αρχέ οικειοποιούνται το όλο εγχείρημα, αλλά έχουμε να κάνουμε με χώρε που βρίσκονται σε κρίση. Οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει είτε στο Μαλί είτε στο Νίγηρα, ε, σε χώρε ε, που έχουν ε, εγγενεί τάσει κρίση μετά την κατάρρευση τη Λιβύη και την διάλυση του Μποκοαράμ και την έλλειψη σταθεροποίηση στο, στο κεντρικό Μαλί δεν υπήρξε κάποια στιγμή έτσι ανακοχής αν θέλετε. Μιλάμε δηλαδή για χώρες οι οποίες είναι ε, εξαιρετικά εύθραυστες, πρέπει να τις υποστηρίξουμε αλλά όχι τυφλά. Υπάρχουν δηλαδή και κάποιες προϋποθέσεις που θέτουμε, κάποιοι όροι και βεβαίως πρέπει να υπάρξει οικειοποίηση σε τοπικό επίπεδο αλλά και ε, να, υπάρξει, να υπάρξουν και ηγετικέ μορφές σε τοπικό επίπεδο. Η διεθνής κοινότητα έχει ε, οργανωθεί κατά αυτόν τον τρόπο G5 Sahel, γιατί ξέρει ότι οι προκλήσει αυτέ που αντιμετωπίζει η περιοχή δεν μπορούν να επιληθούν από ε, μία χώρα ξεχωριστά. Υπάρχουν πολλά διασυνοριακά κοινά προβλήματα, διμερό, τριμερό, ε, κοινά προβλήματα και για των πέντε χωρών και έπρεπε να καθοριστεί πρώτα ένα πολιτικό πλαίσιο εντός του οποίου, και επικοινωνιακό πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Και βεβαίω ε, θα πρέπει μετά αυτό το πλαίσιο να υλοποιηθεί. Ε, είναι λίγο όμως ε, και σαν βαρέλι χωρίς πάτο αυτό, διότι είναι πολλά τα μέτωπα. Ε, οι δομές διακυβέρνησης στις χώρες αυτές δεν είναι και πλέον προσαρμοσμένες στον πληθυσμό τους, ε, στους κινδύνους ασφαλείας, στους δημογραφικούς κινδύνους, στους επιστηστικούς κινδύνους είναι εξαιρετικά περίπλοκο το πρόβλημα. Και θέλουμε να ορίσουμε από κοινού έναν οδικό χάρτη για να προχωρήσουμε, γνωρίζοντας βεβαίως ότι, ότι αυτοί είναι κυρίως που θα πρέπει να οργανώσουν τη δομή της χώρας τους αύριο. Αυτά μπορώ να πω επ' αυτού τώρα. κατά πόσο είμαστε εμείς στη θέση του οδηγού ή όχι. Όχι. Εμείς δίνουμε μια όθηση. Εμείς συνοδεύουμε αυτή τη διαδικασία όσο, γίνει, όσο μπορούμε καλύτερα. Ο κίνδυνος είναι να μην μιλάμε για πλήρη εξάρτηση διότι αλλιώ δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την περιοχή έτσι ώστε τα προβλήματα σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο να εκλείψουν. Τα προβλήματα όμως ισορεύονται αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια απειλή απέναντί μας ε, στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Προσαρμόζεται αυτή η απειλή και βεβαίως εκμεταλλεύεται και τα κενά που έχουν προκύψει είτε λόγω έλλειψης επένδυσης, λίγο, είτε λόγω έλλειψης πολιτικής, ε, ε πολιτικού οράματος ε, και διορατικότητας. Ε, και εδώ είναι που χρειάζεται συνδρομή. Συνδρομή όμως. Έγινε και ένα ερώτημα για τα προγράμματα CBSD Capacity Building for Security and Defense, δημιουργία δυνατοτήτων για την άμυνα και την ασφάλεια. Ε, για να μπορέσουμε, να μπορέσουμε να καλύψουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον εξοπλισμό σε αισθήματα ασφαλείας. Ε, ε, στο Μαλί, παραδείγματος χάρη, ε, για την προστασία του αεροδρομίου, ε, για τη δημιουργία ενός ιατρικού κέντρου και εκεί βοηθάμε. Είναι πολλά τα διδάγματα από τα εγχειρήματα αυτά. Πάντως αυτά, αυτές οι δομές υπάρχουν πλέον σήμερα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό πλαίσιο και τις ασκήσεις που γίνονται, τις στρατιωτικές, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά το ερώτημά σας. Ε, αυτό που θέλουμε είναι οι λόγοι για τους οποίους το Μαλή εχθές ή κάποια άλλες χώρες αύριο ε, καταραίουν να μην ε, εμφανιστούν ξανά. Η δομή ασφάλειας και άμυνας των αφρικανικών χωρών του G5 μιλάω για αυτές τις χώρες και αφήνω και το Τσάτ και τη Μαυριτανία στην άκρη δυσκολεύονται ιδιαίτερα λοιπόν αυτές οι χώρες να αντιμετωπίσουν όλες αυτές, όλες αυτές τις προκλήσεις. Και το G5 είναι πιστεύουμε η σωστή οδός ε, για την ε, αλλαγή αυτή. Μιλάμε για 5.000 άτομα έτσι στο G5 αυτή τη στιγμή, δεν μιλάμε για κάποια τεράστια δύναμη, αλλά θα ασχοληθεί με τις περιοχές που δεν ελέγχονται αυτή τη στιγμή. Ξέρετε ότι σήμερα δεν υπάρχει έννοια των συνόρων για τους, ε, για τις παραμεθόριες, τους παραμεθόριους πληθυσμούς. Έχουμε, μιλάμε για ζώνες οι οποίες δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο και εκεί βεβαίως αυτό ευνοεί το λαθρεμπόριο, ότι δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου. Αναφέρθηκα προηγουμένω στη συμφωνία μεταξύ Τσάντ, του Τσάντ και των γειτονικών χωρών για το δικαίωμα καταδίωξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, ε, αυτές ε, οι οάσεις, έτσι, αυτά τα, οι οάσεις για τους λαθρεμπόρους, εκεί όπου δεν μπορεί να τους κυνηγήσει κανείς, θα εκλείψουν. Ενδεχομένως να μην κατάλαβα καλά το ερώτημά σας, αλλά εμείς τους δίνουμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές και από εκεί πέρα πρέπει να τις εφαρμόσουν αυτοί. Τους βοηθούμε να τις εφαρμόσουν. Διότι εμείς σε επίπεδο και άμυνας δεν κάνουμε κάποια συνοδευτική δράση. Δεν το θέλουν τα κράτη-μέλη άλλωστε. Η συνοδευτική δράση γίνεται είτε από τη Μινουσκά, είτε από την Μπάρκαν, είτε από άλλους ε, παράγοντε από άλλε χώρε. Εμεί κάνουμε, εμείς εργαζόμαστε πλαίσια δημιουργία δυνατοτήτων, capacity building. Ενδεχομένω όμω να το χαρακτηρίσει αυτό και ε, άσκηση και ε, κατάρτιση. Αλλά είπα προηγουμένω στην παρουσίασή μου, το χειρότερο, μου, το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε πράγματα τα οποία γίνονται ήδη. Η ζήτηση υπάρχει μεγάλη. Αναφερθήκατε και εσεί στο συντονισμό. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τι επικαλύψει ή να κάνουμε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα αποδειχθούν άχρηστα. Και για το τελευταίο ερώτημά σα για τη χρηματοδότηση των δημοκρατικών ομάδων. Αυτό είναι ζήτημα ουσίας. Όλοι έχουν ακούσει για τις απαγωγέ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι πάντα δημοκρατικές ομάδες που κάνουν τις απαγωγέ. Μπορεί να είναι μια μορφή επιχείρηση. Έτσι. Κάποιοι ειδικεύονται στι απαγωγέ κάποιοι άλλοι ε, στην ανταλλαγή ε, ομήρων, άλλοι στην διαπραγμάτευση. Όταν βλέπει λοιπόν κανείς τι γίνεται στο μαλλί με τις ε, ΜΚΟ, αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι η απαγωγή ενός ε, δυτικού ε, στο ΣΑΕΛ είναι ένα, ζήτημα, ένα εθνικό ζήτημα και δεν θέλουμε σε κανένα περίπτωση να τροφοδοτήσουμε αυτή τη χρηματοδότηση. Τώρα η οδός της χρηματοδότησης είναι διαβλή. Η χρηματοδότηση είναι περίπλοκη, η σχέση με το οργανωμένο έγκλημα δηλαδή. Ε, υπάρχει αυτή η σχέση. Τώρα πώς θα μπορέσουμε εμείς αυτό να το καλουπώσουμε και να το ελέγξουμε ε, ε, δίνοντας τις εν λόγω χώρες τα μέσα για να μπορέσουν να δράσουν σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου στο ε, σύνολο του εδάφους τους. Βεβαίως αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά για να γίνει χρειάζονται πάρα, πάρα πολλές δράσεις, πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και επανέρχομαι στη δύναμη του G5 και σε αυτές τις περιοχές ε, εκτός ελέγχου, όπου οι τοπικοί πληθυσμοί πραγματικά υποφέρουν, ε, έχουν ξεχάσει τι είναι κράτος, και δείχνει τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς με τη στήριξη στο G5. Ε, μοιραζόμαστε πληροφορίες, δημιουργία, ε, δυνατότητα αντίδρασης μάλλον, δικαστικές διαδικασίε διαδικασίες και δημιουργία δυνατοτήτων έτσι ώστε οι χώρες να συντονιστούν καλύτερα ε, για διασυνοριακά προβλήματα που προκύπτουν. Αυτό κάνουμε στο πλαίσιο του G5. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και όλα τα προγράμματα ανάπτυξης. Ε, έχουμε μια σειρά από δράσει συντονισμένες που αυτή τη στιγμή ακολουθούν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πορεία, δύσκολη βέβαια. Εγώ καθημερινά βλέπω αυτούς που εργάζονται από αυτών των συστημάτων εδώ από τις Βρυξέλλες. Είναι κάτι το οποίο παίρνει πολύ χρόνο και είναι και πολύ δύσκολο να μπορέσει να παρακολουθήσει κανείς δηλαδή το σύνολο της αλυσίδας αυτής. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα ε, την, ε, στα 5 εκατομμύρια που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ειρήνη, 50 αρχικά, 50 μετά, 100 συνολικά. Η Κομισιόν το παρακολουθεί αυτό στενά το συγκεκριμένο κονδύλιο και πώ διατίθεται, διότι υπάρχει μια εταιρική σχέση εντό εισαγωγικών ε, αξιοπιστίας με τις χώρες που υποστηρίζουμε. Πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ε, στην, από την πλευρά του δικαιούχου ε, ότι πρέπει να κάνει και αυτός ε, σωστή δουλειά έτσι ώστε να είναι βιώσιμη αυτή η συνεργασία και όχι εφήμερη. Το G5 που έχει μια, ένα αντίστοιχο προπολογισμό, παραδείγματο χάρη, αυτό είναι κάτι που βοηθάει. Και έρχομαι τώρα στο θέμα του κατά πόσο εμείς είμαστε αυτοί που σπρώχνουν ή ε, αν αυτοί είναι που ελέγχουν την κατάσταση που είναι στη θέση του οδηγού, είναι και αυτό μέρο των βαλίστων πρακτικών που προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε. Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και G5 στον τομέα αυτών. Ε, νομίζω ότι απάντησα στα ερωτήματα, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι. Α, και το τελευταίο, για το European Peace Facility, ε, αργεί ακόμα αυτό, αργεί. Διότι ήταν το πρώτο σας ερώτημα, νομίζω. It was indeed, and thank you for... Αυτή ήταν η τελευταία. Σας ευχαριστώ που την αναφέρατε και αυτή. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ερωτήσεις θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπενουά και εδώ κάθε επιπλέον πληροφορία που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο την πρωτοβουλία για την ειρήνη την αναμένουμε με ενδιαφέρον. Κύριε Μπενουά έχετε το λόγο. Λέγομαι Μπενουά Λότ, εργάζομαι στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Μονάδα Ασφάλεια και Σφαιρικές Απειλές. Θα αναφερθώ στο ερώτημα το σχετικό με τα οικονομικά μέσα που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκαμε στο CDSD και στην διευκόλυνση για την ειρήνη. Ασφάλεια λοιπόν και ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο έχει κινητοποιηθεί όχι υπέρ του G5 γιατί το G5 δημιουργήθηκε πρόσφατα και για την στήριξη του G5 υπάρχει έτσι και αλλιώ το καταπίστευμα για την ειρήνη στην Αφρική ενώ το προηγούμενο δεν μπορεί να κινητοποιηθεί. Μπορεί όμως να κινητοποιηθεί για την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων μεμονωμένα των χωρών των G5 στον βαθμό που έχουν συντονίσει τις δράσεις τους με αναπτυξιακό κατά βάθος στόχο. Έχουν υπάρξει κάποια προγράμματα που έχουν ξεκινήσει ήδη στο Μαλί και άλλα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν περαιτέρω υπέρ των ενόπλων δυνάμεων μεμονωμένα και όχι του δύναμη συνεργασίας. Σχετικά τώρα με την Ευρωπαϊκή Μονάδα, πρωτοβουλία μάλλον για την ειρήνη, θα μπορούσε να κινητοποιηθεί για το G5 γιατί γιατί έχει έτσι και αλλιώ την δυνατότητα να ξεπεράσει ακόμα και τα σύνορα της Αφρικανικής Υπήρου. Αν λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνει δεκτή, τότε θα μπορούσε να υποστηριχθεί από την Επιτροπή το G5 Sahel. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα δούμε αυτά, πώς θα ξεκινήσει η συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας για το συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φραντά για την παρουσία του εδώ και για τα συνολικά σχόλια και παρατηρήσεις που έκανε για την Σαχάρα, για την ομάδα των πέντε. Να ευχαριστήσω επίσης και τον κύριο ε, Μπενουά. Είστε ελεύθεροι. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ λοιπόν. Κλείνουμε το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Θα περάσω τώρα να δώσω τον ρόλο μου ως πρόεδρος και να δώσω την Προεδρία στον κύριο Στέτινα για το 5 και Κυρίε Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γιάρομιρ Στέτινα, λέγομαι. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών και Αντιπρόεδρος της ΣΕΝΤΕ. Η ε, Επιτροπή μας ε, τώρα θα περάσω στο επόμενο θέμα. Και θα ήθελα τώρα να χρησιμοποιήσω την τσεχική. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Οπότε. Έχουμε στην ημερήσια διάταξη τις λεγόμενες υβριδικές άπειλες στην στρατηγική επικοινωνία και θα συζητήσουμε τα θέματα αυτά με την Σίλβια Κάιντς Χούμπερ πρώτα απ' όλα. Καλώς ήρθατε και έχετε τον λόγο. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω την μητρική μου γλώσσα Θα μιλήσω αγγλικά. Καλησπέρα σας. Τώρα θα ήθελα να σας παρουσιάσω μια εικόνα του πακέτου για τις υβριδικές απειλές που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο τέλος Ιουνίου. Το πακέτο πράγματι ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία ζήτησε τον Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή να οικοδομηθεί αντοχή στις υβριδικές απειλές, ειδικά μετά την χημική επίθεση στο Σόλσβερι στην Αγγλία και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μίλησαν για αυξημένη αντοχή σε ραδιοβιοχημικό πόλεμο και τέτοιες απειλές και από την άλλη στην αύξηση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης υβριδικών απειλών όπως κυβερνοπολέμους, στρατηγικές τηλεπικοινωνίες και αντικατασκοπία. Αυτό το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα πακέτο τριών εγγράφων, μία ανακοίνωση που συγκεκριμένα απαντάει στα αιτήματα του Συμβουλίου του Μαρτίου για το πώς μπορούμε να προχωρήσει το θέμα στους πέντε τομείς που ανέφερα. Είχαμε δύο εκθέσεις. Μία έκθεση για την εφαρμογή του κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση και υβριδικών απειλών και η δεκατη η έκθεση για τη γνήσια και αποτελεσματική Ένωση Ασφαλείας. Πριν περάσω στα κύρια μηνύματα, να αναφέρω κάποια γενικά μηνύματα για τις υβριδικές ε, απειλές οι οποίες μας απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν διαφορές δράσεις και πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. Η Κομισιόν και η Πατή Εκπρόσωπος έχουν κάνει πολλές προσπάθειες για να αυξηθούν οι δυνατότητες της Ένωσης για να αντιμετωπίσει ρόβι ταχύ απειλές και υβριδικές απειλές και έχουμε αυτά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς. Έχουμε επίσης διάφορα πλαίσια πολιτικής στα οποία απαιτείται συγκεκριμένη δράση και ένα νέο πλαίσιο πολιτικής επίσης ε, διαμορφώνεται αυτή την στιγμή. Πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Η βασική ευθύνη για την ενίσχυση της αντοχής σε αυτές τις ε, και την ενίσχυση των δυνατοτήτων ε, είναι και θα παραμείνει κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν μπορεί και θα χρησιμοποιήσει τις αρμοδιότητες που έχει για να στηρίξει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειές του, αλλά και πάλι είναι ευθύνη των κρατών μελών. Στην ε, ανακοίνωση αυτή συνοψίζονται τα κυριότερα επιτεύγματα και κυρίως μιλάμε για την πρόοδο που γίνεται και τα κυριότερα έργα στην στρατηγική επικοινωνία και έχουμε τώρα μία ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης ε, που εγκρίστηκε βεβαίως νωρίτερα φέτος, αλλά αυτά θα τα αφήσω να τα πει ο συνάδελφος που θα μπορεί να μας πει πολύ περισσότερα για την αντίληψη του περιβάλλοντος ε, και πάλι υπάρχει μία πλατφόρμα ακριβώ για την αύξηση αυτής της αντίληψης που είναι μια βασική πτυχή αντιμετώπισης των ευρετικών απειλών. Ήταν ένας πυρήνας ο οποίος έχει συσταθεί εντός του ε, και πύχ ε, της ε, εξωτερικής δράσης από το 2016 και μέχρι στιγμής έχει κάνει πάνω από 100 αξιολογήσεις και ενημερώσεις αλλά και πάλι αυτά θα μας τα πει ο εκπρόσωπος εδώ της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το κέντρο αυτό υβριδικών απειλών για την ενίσχυση της ε, αντοχής ειδικά απέναντι σε απειλές ε, ρόβι ταχύ πολέμου θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του τι έχει γίνει τους τελευταίους έξι μήνες δηλαδή μια ανάλυση των κενών ε, της ετοιμότητας για περιστατικά που έχει γίνει τώρα που έχει γίνει και τη μοιραζόμαστε με τα κράτη-μέλη ακριβώς για να αντιληφθούμε πού είναι τα κενά, ποια είναι τα προβλήματα και τι πρέπει να γίνει. Για την ε, δυνατότητα αντίδρασης ε, σε κρίσεις έχουμε την επικοινωνία με τον ΝΑΤΟ που έχει αυξηθεί σημαντικά κυρίως μέσω της ε, άσκηση, της παράλληλης και συντονισμένης άσκησης ε, με ένα σενάριο ευρυδικής απειλής που έγινε για πρώτη φορά το φθηνό που μας πέρασε σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει τις ε, δυνατότητες της για υβριδικές απειλές μεγάλης κλίμακας. Το παράδειγμα αυτό και βέβαια μπορώ να φέρω ε, ε, κάποια παραδείγματα, δείχνουν επίσης, ε, πέρα από την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ότι το πλαίσιο πολιτικής που έχουμε διαμορφώσει και στο οποίο οι δραστηριότητες αυτές έχουν ξεκινήσει, είναι ένα πλαίσιο το οποίο λειτουργεί και αποδίδει και εδώ πέρα αναφέρομαι κυρίως στο κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ξεκίνησε το 2016 με τις 22 δράσεις για την ε, αύξηση της αντοχής, ε, την προετοιμασία και την αντίδραση στις υβριδικές απειλές. Εδώ πέρα αναφέρομαι κυρίως στο σχέδιο δράσης του 2017 με κυριότερο στοιχείο την οδηγία για την ασφάλεια δικτύων ε, και συστημάτων πληροφορικής, η οδηγία ένιση. Επίσης αναφέρομαι στο σχέδιο δράσης ε, Ροβιταχή του 2016 με τα 23 μέτρα και δράσεις και τέλος θα ήθελα να επισημάνω την διακήρυξη της Βαρσοβίας του 2016 που καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΝΑΤΟ Και βεβαίως ε, τα 70 μέτρα που προτείνονται για αυξημένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ που προτείνονται εκεί που αφορούν ζητήματα ευρετικών απειλών. Η κοινή ανακοίνωση επίσης ε, αναφέρει μόνο το τι μπορεί να, τι έχει γίνει και ποια είναι τα μεγάλα επιτεύγματα. αλλά ακριβώς υπάρχει και το ζήτημα των συνεισφορών για την αντιμετώπιση των οροβιταχή επιλών και εδώ πέρα ακριβώς τονίζονται οι... τα κενά που αναφέρονται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ στα όσα είπε ε, λέει η ανακοίνωση αυτή, δηλαδή πώς θα προχωρήσουμε ακριβώς το θέμα της στρατηγικής επικοινωνίας. Υπάρχουν ειδικοί από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που μπορούν να τα εξηγήσουν αυτά. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε άλλους ε, τομείς που ήταν ε, το θέμα των επόμενων βημάτων σε αυτήν την κατεύθυνση και αφορούν ακριβώς την ενίσχυση των δράσεων σε αυτόν τον τομέα. όπου τα μέτρα αυτά ακριβώς ε, έχουν στόχο το πώς θα σεβαστούμε καλύτερα τους διεθνείς κανόνες που υπάρχουν, πώς θα αυξηθεί η αντοχή μας και πώς θα προωθηθεί ακριβώς καλύτερα ο συντονισμός όσον αφορά την άξιση της αντοχής και της αποτροπής στον τομέα αυτόν. Η ανακοίνωση τονίζει την ανησυχία που υπάρχει κυρίως για την εφαρμογή του σχεδίου δράση για την κυβερνοσφάλεια που υπάρχει ήδη και εδώ πέρα ακριβώς ε, ε, επιστήσαμε την προσοχή στο ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με βάση το σχέδιο που είχαμε, δηλαδή μια σύσταση για μια συντονισμένη απάντηση σε περιστατικά κυβερνοπολέμων, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα επίσης το λεγόμενο κουτί της κυβερνοδιπλωματίας ε, και τέλος το ψηφιακό πρόγραμμα που υιοθέτησε η Κομισιόν στις 6 Ιουνίου πριν από 15 μέρες για τον επόμενο κοινοτικό προπολογισμό μετά το 2021. Τέλος, η αύξηση της αντοχής. Και εδώ πέρα να σας δώσω ένα παράδειγμα του τι συζητήθηκε τι ακριβώς θα κάνουμε, γιατί η πρόταση είναι ήδη επιτάπητος, αναφέρομαι στις άμεσες ξένες επενδύσεις από τα κράτη-μέλη και τον ελεγχό τους, πρόταση που ενέκρινε η Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2017 και ελπίζουμε να εγκριθεί γρήγορα από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Να αναφέρω κάποια πράγματα και για την έκθεση προόδου για τις υβριδικές απειλές. Είναι ήδη η δεύτερη έκθεση που ε, έχουμε παρουσιάσει από την έγκριση του πλαισίου το 2016. Έχουμε εδώ πέρα μόνο τα όσα συνέβησαν από την τελευταία έκθεση. Ε, κατά βάση δηλαδή, ένα έτος από πέρσι τον ε, Ιούλιο και τα ανέφερα, μιλάμε για 22 δράσεις, οπότε δεν θέλω και δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα αυτά. Να αναφέρω λοιπόν τρία μηνύματα που προέκυψαν όσον αφορά την αντίληψη του περιβάλλοντος ή της ε, κατάστασης. Έχουμε τώρα όλα εκείνα τα μέσα μα μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε τις υβριδικές απειλέ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ο πυρήνα που ανέφερα ήδη εντός της ΕΕΔ και περιλαμβάνει και στρατιωτικούς ειδικού και μη. Συμμετέχουν εκεί 26 κράτη-μέλη που μέσω αυτού του δικτύου έχουν μια πλατφόρμα ανάλυσης στοιχείων. Το δεύτερο θέμα αφορά ακριβώς ε, το πλασίο του Ελσίνκη. Έχουμε τώρα 15 χώρες που συμμετέχουν εκεί και μοιράζονται την εμπειρία τους στην αντιμετώπιση υβριδικών απειλών. Όσον αφορά την αύξηση της ανθεκτικότητας, ένα βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, απαιτεί δράση σε πολλούς τομείς ε, πολιτικής και αφορά ακριβώς ε, προστασία των κρίσιμων υποδομών, ασφάλεια παροχής. Ε, δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι δράσεις απαραίτητος ε, αφορούν τη συγκεκριμένη απειλή, αλλά θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι θα είναι πιο ανθεκτική η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση τέτοιων απλών. Αυτό το οποίο λοιπόν δείχνει η έκθεση, χωρί να μπω σε πολλέ λεπτομέρειε, είναι ότι έχει σημειωθεί πρόοδο σε όλους τους τομείς πολιτικής ε, που αφορούν αυτό το ζήτημα. Ένα παράδειγμα, η άσκηση καμήρα στον τομέα της υγείας που ελέγχει ακριβώς την προετοιμασία σε περίπτωση επιδημιών και επιπλέον είχαμε και άλλα μέτρα καταπολέμησης της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, ε, της ριζοσπαστικοποίησης και συνεργαζόμαστε και με τον κλάδο για να κατεβαίνει η ρητορική μίσους ε, γρήγορα όταν ανοιχνεύεται. Και τέλος, για την πρόληψη και την αντίδραση, μια καλή περσινή καινοτομία ήταν για πρώτη φορά η παράλληλη και συντονισμένη άσκηση τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ΝΑΤΟ για να δούμε τις ε, δυνατότητές μας με βάση συγκεκριμένα σενάρια για το πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε υβριδικές απειλές. Τελευταία λέξη για την ε, συνεργασία με το ΝΑΤΟ που προφανώς είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο σε οτιδήποτε κάνουμε για τις υβριδικές απειλές. Ανέφερα ήδη το κοινό πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, ένα πλαίσιο πολιτικής για συνεργασία με τον ΝΑΤΟ στον τομέα από τις 74 ε, αυτές ε, δράσεις που ήδη από αυτές οι 20 εστιάζουν στις υβριδικές απειλές και πάλι έχουμε εδώ πέρα κάποια βασικά στοιχεία Έχουμε τον πυρήνα, έχουμε τον αρμόδιο κλάδο του ΝΑΤΟ και το κέντρο αριστείας στο Ελσίνκι που είναι σε τακτική επαφή μεταξύ τους και έχουν ε, σχέσεις ε, εργασίας και τώρα προσπαθούν ακριβώς ε, να προχωρήσουν σε μια τριμερή συνεργασία με υλικό από ανοιχτές πηγές. Το κέντρο αριστείας έχει στόχο να στηρίξει το προσωπικό της Ένωσης και του ΝΑΤΟ που εργάζεται σε τέτοιες απειλές Μιλάμε για εργαστήρια, ασκήσεις, σεμινάρια για να αντιληφθούμε την φύση των υβριδικών απειλών και ένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα του τύπου των εργαστηριών που θα οργανωθούν παραδείγματος χάρη το πιο πρόσφατο σενάριο αφορά ακριβώς ε, τις συνθήκες ε, υβριδικής απειλής και τέλος έχουμε τις επαφές του προσωπικού που προβλέπει η κοινή δήλωση, οι οποίοι συνεχίζονται σε πολλούς τομείς. Και βεβαίως είχαμε ακριβώς πλέον αύξηση και των επαφών, του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων. Λοιπόν, τα έγγραφα δείχνουν και δεν έχω μπει ακόμα σε πολλές λεπτομέρειες ότι πολλά πράγματα έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι λειτουργούν δείχνει ότι έχουμε τις πρώτες δραστηριότητες και ότι αυτό το οποίο πραγματικά είναι απολύτως απαραίτητο ναι είναι η ενημέρωση αφενός η σαφής εικόνα αλλά είναι η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας και τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Λοιπόν, θα μιλήσω τώρα τη μητρική μου γλώσσα, τα τσεχικά. καλό απόγευμα στους συναδέλφους και τον κύριο Ζιλ Πόρτμαν, τον team leader της Task Force από την Υπηρεσία εξωτερική Δράσης. καθώς και τον Κάβορη Κλόντι, τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Προγραμματισμού πάλι στην υπηρεσία εξωτερικής Συνεχίζω στα τσεχικά. Ε, αξιοτιμική έχετε το λόγο. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο πρώτος. Ο κύριο Σικλόντι, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε και συγγνώμη που άργησα κάπως για να έρθω σε αυτό το πάνελ. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια χωρίς να επαναλάβω αυτά που είπε και που εξήγησε ήδη η Σίλβια. Δύο λόγια για το ε, τοπίο στο τεφρά αφορά τις απειλές το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση. Δεν έχει αλλάξει το υβριδικό τοπίο απειλή ε, Σίγουρα δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Υπάρχουν κυβερνοδραστηριότητε, ε, κυβερνοαπειλές ε, των κρίσιμων υποδομών μας, των συστημάτων μας, παραπληροφόρηση, ολόκληρε εκστρατείε παραπληροφόρησης. Ορισμένε φορές έχουμε και εξαιρετικά εχθρικές επιθετικές στρατιωτικές δράσεις ε, κοντά στα σύνορά μας. Ο σκοπός είναι πάντα ο ίδιος. Η αποσταθεροποίηση των χωρών μας, των κοινωνιών μας, να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη του, της κοινής νόμης προς την κυβέρνηση, προς τους θεσμούς ε, και να βεβαίως να δουν, να δοκιμάσουν ποια είναι η δυνατότητα αντίδρασης, απάντησης. Και βεβαίως είχαμε το Σόσμπορι, ε, που μας ε, θύμισε την πραγματικότητα, τι μπορεί να συμβεί στο, στο έδαφος της Ένωσης, ότι μπορεί να γίνουν τέτοιες περικαλαιότητες, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Αφενός ένας στόχος είναι να εντοπίζουμε όσο γίνεται πιο νωρίς αυτές τις ε, δραστηριότητες πριν λάβουν χώρα οι δράσεις. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάποια γεγονότα που μοιάζουν απομονωμένα ορισμένε φορές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερη καμπάνιας, μιας ευρύτερη εκστρατείας. Εξού και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά ε, μετατρέπονται σε υβριδική δραστηριότητα και βεβαίω πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί για να μπορούν οι κοινωνίες μας, οι υποδομές μας, οι θεσμοί μας να μπορούν ε, να ε, αντέξουν απέναντι σε μια τέτοια επίθεση, να μην είμαστε ευάλωτοι απέναντι σε τέτοιε επιθέσεις. Για να συμβεί αυτό πρέπει να καταλάβουμε ε, ποια είναι τα κρίσιμα ε, σημεία, ε, τα ευάλωτα, για να μειωθούν τα ευάλωτα αυτά σημεία. Είναι βεβαίως ένα ζήτημα εθνικής αρμοδιότητας πρωτίστως, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει μια χρήσιμη πλατφόρμα για να ενισχύσει αυτέ τι εθνικέ προσπάθειε για να επιτευχθούν τα αποτελέσματα. Μια σωστή ανθεκτικότητα σημαίνει ε, να υπάρχει και μια σωστή δύναμη αποτροπή. Ε, στέλνουμε δηλαδή το μήνυμα ότι θα δυσκολευτεί όποιο θελήσει να μα επιτεθεί. Πρέπει επίση να συντονίσουμε την απάντησή μα απέναντι σε τέτοιου είδου υβριδικέ ε, δραστηριότητε. Θα πρέπει να έχουμε του κατάλληλου μηχανισμού απόκριση για να μπορούμε γρήγορα και αποτελεσματικά να συντονιστούμε και να υποστηρίξουμε τη χώρα που έχει ε, υποστεί την επίθεση. Πρέπει να συνεργαστούμε στα πλαίσια των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, με το ΝΑΤΟ, ε, να υπάρχει μια ε, διακυβερνητική προσέγγιση. Συχνά ε, οι υβριδικές πτές επιθέσεις ε, είναι εκτός αυτής της σφαιρικής προσέγγισης. Η απάντησή μας μπορεί να είναι επιτυχημένη μόνο να συντονιστούμε μεταξύ κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά την απάντηση απέναντι σε τέτοιου δραστηριότητε. Επίση, θα πρέπει να, να ε, κινητοποιήσουμε τη βιομηχανία αλλά και την κοινωνία, το σύνολο της κοινωνίας ε, θα πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένο για να έχουμε μια σωστή απάντηση. Και τέλος, στο πλαίσιο αυτό να πω ότι όπως θα γνωρίζετε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την αντιμετώπιση των ευρυδικών απειλών και την αύξηση της ανθεκτικότητας δεν επικεντρώνεται μόνο στα κράτη-μέλη, αλλά και στις εταιρικέ χώρες, στις χώρες εταίρους, συγγνώμη τις γειτονικέ μας χώρες. Εμείς επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στην κοινή ε, ανακοίνωση που έχει προετοιμαστεί και θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Σύλβια ε, Σίλβια αναφέρθηκε σε αυτό η Σίλβια λεπτομερώς είμαι βέβαιος. Ε, στο Μάρτιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου και μετά τα γεγονότα του Σόλσμπερι ελέγχθη ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πρώτης μέγιστης ανησυχίας. Θα πρέπει να δούμε ε, λοιπόν ποιες δράσεις μπορούμε να αναλάβουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των χωρών μας και των κοινωνιών μας. Τρία έγγραφα λοιπόν ε, εκπονήθηκαν με σκοπό την ενίσχυση του ίδιου ακριβώς μηνύματος. Έχουμε μια κοινή ανακοίνωση Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τη ΥΠΑ της εκπροσώπου, όπως ζητήθηκε από το Μάρτιο του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό βεβαίως φτάνει και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο. Η κοινή ανακοίνωση έχει ως σκοπό να προσανατολίζεται προς συγκεκριμένε δράσεις, δηλαδή να εντοπίσουμε συγκεκριμένα βήματα μέσα των οποίων μπορούμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορεί να απαντήσει σε τέτοιου είδους υβριδικές ε, δράσεις. Ε, υπάρχει και ένα κοινό πλαίσιο, το ανέφερε η Σίλβια, είναι η απάντηση στα 22 σημεία δράσης, είναι, έχουμε τη δεύτερη ετήσια έκθεση από αυτού. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μέσω αυτού, ε, έτσι με ένα σφαιρικό τρόπο, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενημερώνουν με διαφάνεια τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά το τι κάνουν, τι έχουν κάνει τα τελευταία έτη κατά την εφαρμογή αυτών των 22 δράσεων. Και υπάρχει και μια έκθεση που είναι αυτό της ε, Task Force για την Ασφάλεια της Ένωσης που επικεντρώνεται κυρίως στο CBRN, στις σχετικές επιθέσεις, αλλά ασχολείται και με μια σειρά ακόμα τομείς μεταξύ των οποίων ε, και οι κυβερνητικές επιθέσεις. Ε, να πω δύο λόγια ακόμα για την κοινή ανακοίνωση επικεντρώνεται σε πέντε τομείς. Ένας από αυτούς είναι η ευαισθητοποίηση και είναι το πιο σημαντικό για να μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, συμβαίνει γύρω μας. Ε, εδώ δίνεται έμφαση σε δύο στοιχεία. Πρώτον, θα πρέπει να εντοπίσουμε οποιαδήποτε ε, βλαβερή δράση το συντομότερο δυνατόν, διότι πρέπει να τις προλάβουμε και όχι να προσπαθούμε να τι αντιμετωπίσουμε των υστέρων. Δεύτερον, να καταλάβουμε πώς συνδέονται μεταξύ τους. Έχει δημιουργηθεί ε, ένα fusion cell για το θέμα αυτό στην υπηρεσία εξωτερική δράση, ε, μια μονάδα που πλέον είναι πλήρω επιχειρησιακή από τον περασμένο Ιούλιο. Ε, οι δυνατότητε τη δοκιμάστηκαν ήδη ε, στις συντονισμένες ασκήσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πέρυσι είχαμε πάνω από 100 προϊόντα που βοηθούν ε, τους ε, λαμβάνοντες τις αποφάσεις ε, στο έργο τους είναι σαφές μετά και το Σόσμπερι και με βάση και την εντολή που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο ότι σε κάποιους τομείς θα πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες δυνατότητες στον τομέα του κυβερνοχώρου CBRN και ε, οι πληροφορίες, πληροφοριών. Είναι τομείς οι οποίοι δεν έχουν, ε, δεν έχουν ε, καλυφθεί επαρκώς, όπου υπάρχει περιθώριο για περισσότερους πόρους για να, για να υπάρξει πρόοδος. είναι επίσης σημαντικό να συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ στα πλαίσια του Fusion Cell και της και του κλάδου της ανάλυσης ε, και να συνεργαστούμε και με το κέντρο αριστείας του Ελσίνκη. Έχουμε διενεργήσει μια μελέτη κινδύνου στα κράτη-μέλη. το η πρώτη δράση στα πλαίσια του κοινού πλαισίου. Αυτό έγινε στα πλαίσια της ομάδας φίλων της Προεδρίας. Θα υποβάλει την έκθεση του ε, στο τέλος του έτους. Ε, χωρίς να ονοματίζουμε, χώρες, ε, αλλά ε, αναφερόμενοι στα πιο, στα πιο ευάλωτα σημεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν και θα πρέπει να, να διορθώσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η εντολή αυτή, η εντολή του μάλλον έχει ε, διευρυνθεί τουλάχιστον στο 2020 για να βοηθήσει τα ευρωπαϊκά σημεία και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει και το κέντρο αριστείας, το οποίο πέρα από την έρευνα πέρα από τις ασκήσεις και τα εργαστήρια για τις χώρες εταίρους μπορεί να αρχίσει να εξετάζει και ορισμένα αρκετά ευαίσθητα ζητήματα όπως τα ευάλωτα σημεία στα κράτη-μέλη με μια πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση να μπορούμε να αναδείξουμε κάποιες από αυτές τις ευάλωτες ε, τα ατεβάλλοντα σημεία. Μπορεί να ασχοληθεί, ασχοληθεί και με άλλα ευαίσθητα ζητήματα, όπω το πώ μπορούν να ενεργοποιηθούν ε, κάποιοι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, όπω το 42,7 ε, ε, για την αμοιβαία συνδρομή, υπό ποιε προποθέσει μπορούν να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα άρθρα και πώς, ποια είναι η διάδραση μεταξύ αυτών των μηχανισμών. Όχι μεταξύ μόνο αυτών των δύο ευρωπαϊκών μηχανισμών, αλλά και του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Μετά, το CBRN, εδώ ο στόχος είναι να έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα έγκαιρα. Αυτό χρειάζεται χρήση σημαντικής δουλειάς σε επίπεδο πληροφοριών. Ε, θα πρέπει να έχουμε δυνατότητες εντοπισμού ε, των ε, ε, λαθρεμπόρων ουσιών, CBRN. Από εκεί πέρα θα πρέπει να υπάρχει και μία θα πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει εφόσον λάβει χώρο με τέτοια επίθεση για να μπορέσει να επανέλθει η ομαλότητα. Ε, να σας πω ότι και στα πλαίσια των μόνιμης δομής ΠΕΣΚΟ υπάρχουν ιδέες μεταξύ και των κρατών μελών για την δημιουργία μιας ε, δύναμης η οποία να μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα και να βοηθήσει. Πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης μια βάση δεδομένων όπου θα υπάρχει ένας κατάλογος όλων των χημικών ουσιών, ε, χημικών δραστικών ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις CBRN. Ε, θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο επίσης ε, υγειονομικών οργανισμών και αρχών που, θα, που μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσουν και να έχουμε και ένα απόθεμα φαρμάκων για να μπορούμε γρήγορα να βοηθήσουμε τη χώρα που θα έχει χτυπηθεί. Θα πρέπει να λάβουν χώρα επίσης ασκήσεις και θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι και οι διεθνείς κανόνες στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχει μια σύμβαση για τα χημικά όπλα με πολύ αυστηρούς κανόνες. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς συμμόρφωσης ε, με τη σύμβαση αυτή και βεβαίως αυτό περιλαμβάνει και την επιβολή κυρώσεων ή χρειαστεί, εφόσον χρειαστεί ε, για να μπορέσουν να αποτραπούν κάποιες χώρες ή κάποιες οργανώσεις από το να χρησιμοποιήσουν ε, επιθέσεις CBRN. Ε, η στρατηγική επικοινωνία είναι ένα θέμα το οποίο θα, και ο Τζάι, θα αναφερθεί ο Τζάι στη συνέχεια. Τώρα για τι κυβερνοεπιθέσει, που είναι ο τέταρτο τομέα Εδώ είναι προφανέ, προφανές ότι μιλάμε για μια κρίσιμη απειλή για τι κοινωνίε μα και τι υποδομέ μα. Έχουμε πολύ καλά εργαλεία στην πρώτα, στην διάθεσή μα στην οδηγία νης που είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας ε, σε κρίσιμους ε, βιομηχανικούς τομείς, ε, την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας που θα ενισχυθεί. Η Σίλβια αναφέρθηκε προηγουμένως στο blueprint για την εργαλειοθήκη κυβερνοδιπλωματίας που αναφέρεται και σε κυρώσεις για όταν χρησιμοποιούνται κάποια κυβερνοεργαλεία για να παρθούν μέτρα και εκεί βεβαίως που προσπαθούμε εμείς να, να δώσουμε έμφαση, να δώσουμε βάρος, είναι να, το τομέα της κατάρτισης, διότι στον συγκεκριμένο τομέα ε, είναι σημαντικό να υπάρχουν εμπειρογνώμονες ε, ε, ειδικοί. Ίσως να είναι και πιο σημαντικό από την ίδια την τεχνολογία. Ε, πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο ε, συνασπισμένο έτσι ώστε να προστατεύσουμε όλους τους θεσμούς μας, όλες τις αποστολές μας, τις επιχειρήσεις μας, τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να υπάρχει λοιπόν μια κοινή ε, παρακολούθηση αυτών των δικτύων και βεβαίως να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ε, στην κατανομή. Αυτό από μόνο του είναι μια πρόκληση και βεβαίως υπάρχει το θέμα των υπηρεσιών πληροφορίας ευαίσθητο το ζήτημα. Ε, είναι ευθύνη των κρατών μελών. Κατά πρώτον, θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν μεταξύ τους ε, περισσότερο για να έχουμε και μια καλύτερη εικόνα του τι είδους δραστηριότητε ε, προσπαθούμε να προσπαθούμε να εστιάσουμε δεν είναι όμω θέμα μόνο συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Πρέπει επίση να προστατεύσουμε του θεσμού μα. Και ειλικρινά, εάν δείτε τι συμβαίνει ε, στα θεσμικά όργανα ευρωπαϊκά, όλα χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία. Και εκεί βεβαίω θα πρέπει οι δυνατότητέ μα ε, να ενισχυθούν. Υπάρχουν ζητήματα όταν παραδείγματο χάρη είναι ε, ε, υπάλληλο ε, των μυστικών υπηρεσιών ε, βρεθεί, εντοπιστεί, θα πρέπει να μην μπορεί να επιχειρήσει σε ένα άλλο κράτο μέλο σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή θα πρέπει εκεί να υπάρξει ένα συντονισμό. Και τέλο, για το κοινό πλαίσιο, δεν θα μπω βέβαια στα 22 σημεία, αλλά να πω δύο, να πω δύο πράγματα. Πρόκειται για ένα έγγραφο δύο ετών. Έτσι, ε, πολλά έχουν γίνει έκτοτε. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εμείς θα εστιάσουμε στα σωστά σημεία και θα επικαιροποιούμε το περιεχόμενο του κοινού πλαισίου. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η στρατιωτική κινητικότητα. Ε, πολύ σημαντικό θέμα. Οι υβριδικές επιθέσεις ε, κατά των διαφόρων διάβλων που δημιουργούνται μέσω της στρατιωτικής κινητικότητας είναι κάτι το οποίο χρήζει προστασίας. Πρέπει δηλαδή ε, να έχουμε συστήματα backup για να εξασφαλίσουμε, να ε, καταστήσουμε ασφαλείς, ασφαλείς αυτούς τους διάβλους. Και τέλος να πω ότι υπάρχει το επιχειρησιακό πρωτόκολλο το οποίο έχουμε αναπτύξει μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που μας επιτρέπει να έχουμε μια γρήγορη και συντονισμένη απάντηση εφόσον μια χώρα δεχθεί απειλή και ζητήσει βοήθεια. Ε, το έχουμε δοκιμάσει αυτό, το δοκιμάσαμε το προηγούμενο φθινόπωρο σε μια άσκηση συντονισμού μας με, την Ευρωπα... με, τον, με τον θα πρέπει και και οι δύο πλευρές όμως και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικαιροποιήσουν αυτό το πρωτόκολλο έτσι ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί ε, όταν χορηγούμε αυτή την υποστήριξη. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πότμαν. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από τρία χρόνια συστήσαμε αυτήν την ομάδα δράσης, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε αναγνωρίσει μία πρόκληση που δεν αναγνωριζόταν όσον αφορά την επικοινωνία μας προς Ανατολάς. Οπότε ε, συστάθηκε αυτή η ομάδα με τρεις στόχους. Πρώτον, να εξηγήσουμε καλύτερα το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους γειτονές της προς Ανατολάς συνεργαστούμε με άλλους για ποιοτικότερα ΜΜΕ στην περιοχή. Και τρίτον, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα αντίδραση στην παραπληροφόρηση του Κρεμλίνου. Αυτά πρέπει να τα δούμε λοιπόν ε, εν συνόλο. Και βεβαίως η δυνατότητα στρατηγικών επικοινωνιών έχει διευρυνθεί. Έχουμε τώρα ομάδες δράσης που καλύπτουν τα Δυτικά Βαλκάνια και την Νότια Γειτονιά. Οπότε οι ηγέτες αναγνώρισαν τότε ότι η εξωτερική παραπληροφόρηση ήταν μια πραγματική απειλή ασφαλείας και έπρεπε να την αντιληφθούμε καλύτερα και νομίζω ότι ε, αναγνώρισαν ξεκάθαρα ότι είναι μέλος μιας ευρύτερης υβριδικής απειλής και αφορά ζητήματα που ανέφεραν ομιλητές, επιθέσεις δηλαδή μεταξύ άλλων, στρατιωτικές απειλέ, αλλά και πράγματα όπως ε, τα τρόλ του διαδικτύου, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Οπότε τώρα μετά από τρία χρόνια έχουμε νομίζω μια καλύτερη αντίληψη των προκλήσεων, μια καλύτερη αντίληψη της παραπληροφόρησης και της στρατηγικής παραπληροφόρησης που έχει πολλές μορφές και εργαλεία και διάβλους. Αλλά βλέπουμε ότι τα βασικά μηνύματα είναι σταθερά, ότι η Ευρώπη καταραίει, είναι ανήθικη, ότι είναι επιθετική, ότι οι σύμμαχοι μας είναι εξτρεμιστές, οι ανύπαρκτοι από την άλλη και ότι οι παράνομες δράσεις ε, άλλων είναι απλά εναλλακτικές ερμηνείες του διεθνούς δικαίου. Οπότε τα τελευταία τρία χρόνια κάθε εβδομάδα συλλέγουμε παραδείγματα παραπληροφόρησης και ε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε γι' αυτά. Αλλά και τα, να τα αναλύσουμε, να δούμε πώς λειτουργεί μια εκστρατεία παραπληροφόρησης, πώς μπορεί να μας υπονομεύσει και έχουμε καταγράψει 4.000 παραδείγματα παραπληροφόρησης Βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα αφηγήματα που επανέρχονται και κάποιες τακτικές που επανέρχονται. Παράδειγμα τους χάρη. Η δηλητηρίαση του Σκρίπαλ στο Σόλσμπερι αναφέρθηκε. Καταγράψαμε 31 τέτοια αφηγήματα, διάφορες ε, θεωρίες ε, συνωμοσία. Ε, ας δούμε τους χάρη την πτήση των μαλαισιανών αερογραμμών. Έχουμε καταγράψει 57 τέτοια παραδείγματα με στόχο να συσκοτήσουν την αλήθεια και να εμποδίσουν τη δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν σαφές ότι υπάρχει παραπληροφόρηση με στόχο να προκαλέσει σύγχυση, να καθυστερήσει τις αντιδράσεις μας, να διαχωρίσει και να διασπάσει, να αγγίξει βεβαίως και να διεγείρει κάποιες ανησυχίες που υπάρχουν στην Ευρώπη αλλά να τις οδηγήσει σε βαθμό υπερβολής ε, να υπονομεύσει την πίστη μας στα κύρια ΜΜΕ και φορείς της πολιτικής και έχουμε τώρα έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό 1,1 ε, εκατομμύρια φέτος, ειδικά για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Για πρώτη φορά έχουμε ειδική γραμμή του προπολογισμού για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και οριστικοποιούμε τώρα τα σχέδιά μας για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συλλέγουμε δεδομένα και να φροντίσουμε η ανάλυση μας να βασίζεται σε αντικειμενικές ε, πληροφορίες ε, και θέλουμε στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε μια πιο επαγγελματική και τεχνική παρακολούθηση του κυβερνού χώρου και να υπάρχει μια ποσοτική και ποιοτική, δηλαδή ποιοτική εννοώ, τακτική επαγγελματική παρακολούθηση των ΜΜΕ και να υπάρχει και ανάλυση μαζικών δεδομένων για να αντιληφθούμε όχι μόνο το μήνυμα αλλά και σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται και το τρίτο ιδεοδός θα είναι να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη του αντικτύπου στο ακροατήριο. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβανόμαστε την πρόθεση, αλλά ο αντίκτυπος είναι κάτι το, είναι, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε χωρίς να υπάρχουν δημοσκοπήσεις και έρευνα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερα δεδομένα, μεγαλύτερη ανάλυση και παράλληλα με αυτά πρέπει να συνεχίσει η ενημέρωση για τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να πολεμήσουμε την ε, παραπληροφόρηση αντιδρώντας ε, σε κάθε συγκεκριμένη ψευδή Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ένα βήμα προς τα πίσω και να δούμε ποιο είναι το νήμα που τα ενώνει, που προσπαθεί δηλαδή να παραπληροφορήσει αντί να πληροφορήσει. Και αν μπορέσουμε έτσι να καταδείξουμε αυτά τα κοινά μοτίβα θα έχουμε και κάποια ανοσία σε μελλοντική παραπληροφόρηση. Και πρέπει επίσης να συντονιζόμαστε πολύ καλύτερα. Και πρέπει ακριβώς να φροντίσουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε να συνεισφέρουν σε αυτή την ευρύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για να συνεισφέρουμε σε αυτό τον ευρύτερο χώρο συζήτησης και βεβαίω να συντονιζόμαστε με τα κράτη-μέλη. Ε, η ευθύνη παραμένει στα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα όριο στο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές και να μοιραστούμε κάποιες καλές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει στα κράτη-μέλη, αλλά από διαφορετικά υπουργεία καμιά φορά και δεν είναι ορατές σε ολόκληρη την Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρότερος ρόλος για την μεταξύ μας επικοινωνία με τα κοινοβούλια, με τα κράτη-μέλη και με τις αντιπροσωπείες της Ένωσης σε ολόκληρη την Ήπειρο για να φροντίσουμε έτσι να έχουμε μια γενικότερη εικόνα των προκλήσεων. Και τέλος, Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για τους πόρους που απαιτούνται για να είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο. Όχι μόνο πόρους προϋπολογισμού που είναι βεβαίως κάτι το πολύ θετικό αλλά και όσον αφορά τον χρόνο και το προσωπικό που απαιτείται ακριβώς για να αντιληφθούμε την απειλή αυτή σε ολόκληρη σας ευχαριστώ κύριε Πόρτμαν. Ε, να ξεκινήσει κάποια συζήτηση εφόσον το επιθυμείτε. Κύριε Γκάλα, έχετε ερωτήσεις. Έπρεπε να χαιρετήσω μια ομάδα επισκεπτών, γι' αυτό λοιπόν για 15 λεπτά μετά από την πρώτη ομιλία δεν άκουσα την αρχή της δικής σας ομιλίας. Θα ήθελα όμως σαν πολιτική παρατήρηση να πω ότι η πολιτική μου ομάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές και θα στηρίξουμε για να υπάρξουν τα επιπλέον χρήματα τα οποία έχει ήδη αποφασιστεί Τουλάχιστον βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε σε θέση βέβαια να γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχει αυτό το θέμα και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε με ικανοποιητικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει. Να εκφράσω την ευχή ότι όταν υπάρξει μια στρατηγική αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών, η στρατηγική αυτή για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας και των ψευδών ειδήσεων δεν είναι νέες ψευδές ειδήσει, αλλά η αλήθεια. Η αλήθεια είναι το πιο πιστικό μέσο. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε ικανές τις κοινωνίες μας να αναπτύξει την δυνατότητα διάκρισης ανάμεσα στα, στις ψευδείς ειδήσει και τις πραγματικές ειδήσει. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες νομίζω ότι και με τα μέσα ενημέρωσης, και με κοινωνικά μέσα δικτύωσης που έχουμε, στο παρελθόν οι τεχνολογίες δεν ήσαν διαθέσιμες Ξέραμε τι ακριβώς γινόταν, ξέραμε τι ήταν η κομμουνιστική προπαγάνδα σαν παράδειγμα και υπήρχε μια πολλαπλότητα απόψεων η οποία επέτρεπε όμως να ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις και ε, ποια ήταν η σωστή πλευρά. Τώρα υπάρχει μια τεράστια ποικιλία απόψεων, δεν υπάρχει πλέον κομμουνιστική προπαγάνδα, αλλά υπάρχουν κάποιες τάσεις πρόκλησης προβλημάτων, ενόχλησης, να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει μία πραγματική αλήθεια, αλλά ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του αλήθεια. Είναι μία πρόκληση αυτό και διαρωτώ με πώς με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τους εμπλεκομένους και όχι μόνον εσάς αλλά και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης να πείσουν το κοινό τους, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα κοινό το οποίο σίγουρα δεν θέλει να υπάρχουν συγκρούσεις και ιδιαίτερα με ισχύρους γείτονες, πώς θα πρέπει ακριβώς να κατανοήσει το κοινό ότι εν πολλής αμφισβητούμεθα και πιεζόμεθα εδώ λοιπόν έχω απορίες, δεν έχω ακόμα ξεκάθαρες απαντήσεις, αλλά όπως είπα το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, να γνωρίζουμε τι είναι ψευδές και τι αληθινό και να εμείνουμε στο αληθινό, όχι μόνο στο δικό μας αληθινό, αλλά στο πραγματικό. Και έτσι θα μπορέσουμε να πείσουμε τους άλλους πολίτες ότι είμαστε καλύτερη πηγή ενημέρωσης από την άλλη πλευρά. Ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά σας. Έχω δύο μιλητές ακόμα και εγώ θα ήθελα να πάρω το λόγο. Ο κύριος Ντόνζο αλλά παίρνει ο κύριος Φρόιν το λόγο. Αν ήταν εδώ η κυρία Κάιντς Χούμπερ φυσικά ε, θα μπορούσα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα πιο εύκολα. Με ενδιαφέρον άκουσα τον Μάικλ Γκάλ διότι πράγματι διαρωτώ με ε, οι λαοί στην Ανατολική Ευρώπη στη δεκαετία του 60 και του 70 όταν άκουγαν τη φωνή της Αμερικής ε, ή το Radio Free Europe Δεν θέλω να μικρύνω τη σημασία αυτού που γίνεται σήμερα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε με τη Ρωσία ένα σοβαρό πρόβλημα σήμερα. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε εμείς κάνει στο παρελθόν, στη δεκαετία του 70 και του 80, δεν ήταν μόνο η αλήθεια την οποία προσπαθήσαμε να διαδώσουμε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Υπήρχε ένας, μια χαλαρότητα to me uh, There's υπάρχει πάντα και η άλλη πλευρά του νομίσματος, αν όχι σήμερα στο παρελθόν. Ε, συγγνώμη για την παρέκβαση αυτή. Και αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι το που βρισκόμαστε σήμερα για ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ για τα θέματα ενέργειας οι βιβλικές απειλές στις ενεργειακές μας υποδομές. Δεν ακούω πολλά γι' αυτό. Αν και όλοι γνωρίζουμε, έχοντας διαβάσει αρκετά βιβλία, ότι ό,τι συμβεί στις υποδομές μας στον τομέα της ενέργειας θα μας επηρεάσει όλους με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανεπανάληπτος. Το θέμα δεν είναι ότι θα σβήσουν τα φώτα, αυτό είναι το πιο απλό να πιστέψει κανείς. Αλλά αυτό το πλαστικό μπουκάλι δεν θα το έχουμε. Δεν θα υπάρχουν επικοινωνίες, δεν θα υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, ε, να μην πω για τα σανσέρ, γιατί έχουμε και τις σκάλες. Πάντως καταλαβαίνετε ότι είμαστε τόσο εξαρτημένοι από τον ηλεκτρισμό και από την ηλεκτρική ενέργεια που ό,τι και αν συμβεί στα κέντρα παραγωγής και διανομής αυτής της ενέργειας στην καθημερινότητά μας θα έχει τρομακτικές συνέπειες στην ίδια αυτή καθημερινότητα. Α, είναι κάτι το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Merci. Ε, Merci de vos interventions. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω δεν είναι κάτι που στρέφεται εναντίον του ίδιου του ομιλητή. Θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος, αλλά πραγματικά νομίζω ότι λέμε πραγματικά πολλές σαχλαμάρες. Όταν μιλάμε για υβριδικές απειλές, α, τεράστιο τομέα. Βάζουμε ό,τι θέλεις κανείς μέσα. Ε, μια επίθεση ε, στον τομέα των χημικό και βιολογικό με χημικούς και βιολογικούς παράγοντες το ξέρουμε εδώ και 30 χρόνια. Οι κυβερνητικές επιθέσεις, οι τρομοκρατικές επίσης είναι τρομοκρατικές οι απειλές στους λιμένες μας ή στα αεροδρόμια μας. Ε, το έχουμε μπροστά μας εδώ και 60 χρόνια. Η παραπληροφόρηση ε, δεν είναι όλα αυτά υβριδικά. Όλα τα βάζουμε αυτά μαζί βέβαια, αλλά δεν είναι υβριδικά, οπότε δεν είναι τίποτα καινούριο. Τα νιώσαμε αυτά και στον ψυχρό πόλεμο. Απειλές στρατηγικές με προπαγάνδα, κατασκοπία, ανατρεπτικές δράσεις, όλα αυτά τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Λοιπόν, εγώ ακούω υβριδικές, υβριδικές, υβριδικές, λες και ξαφνικά ανακαλύψαμε ε, την αρχή του κόσμου. Εντάξει, στην Κρυμαία υπήρξαν τέτοιου είδους ενέργειες, αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί είμαστε τόσο κολλημένοι σήμερα. Έχουμε πυρηνικές μονάδες παραγωγής εδώ και 40 χρόνια. 40 χρόνια σκεφτόμαστε την ασφάλειά τους και σε επίπεδο πληροφορικό χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να σχεδιάζουμε ένα σχέδιο για την υβριδική απειλή. Ε, πρέπει να είμαστε, ε, να σεβόμαστε την πραγματικότητα. Ε, τα fake news, οι ψευδείς ειδήσει. Προπαγάνδα είναι αυτή. Γιατί να δώσω εκατομμύρια εγώ για να φτιάξω μία μονάδα στις Βρυξέλλες για να διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος. Κοιτάξτε, εγώ να σας πω ότι όταν κάποιος πιστεύει κάτι δεν του το βγάζετε από το κεφάλι τα κέντρα της προπαγάνδας δεν είναι μόνο στο Κρεμλίνο, είναι στο σπίτι μας, είναι στις κυβερνήσεις μας. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ιταλία. Στην ουσία δηλαδή χάρη σε ένα πυρήνα στις Βρυξέλλες θα <coughs> προσπαθήσουμε να περάσουμε στην απομόλυνση αυτών οι οποίοι γεννούν τις ψευδείς ειδήσει. Όχι, πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Είναι άχρηστο κάτι τέτοιο. Μιλάμε για ένα πόλεμο ιδεών, για ένα ιδεολογικό πόλεμο με τα μέσα της πυθούς, με τα μέσα της αλήθειας, με τα μέσα της πολιτικής, αλλά τώρα να βγάψουμε μια υπηρεσία που θα διακρίνει την αλήθεια από το ψεύδος είναι εντελώς λάθος. Και ταυτόχρονα σε όλες τις ε, σε όλες τις, ε, σε όλους τους αρχισυντάκτες και τα λοιπά, στις εφημερίδες και τα λοιπά, στα κανάλια, σε εφημερίδες μεγάλες όπως το Μόντο και τα λοιπά. Όλα αυτά επηρεάζουν τον κόσμο πολύ περισσότερο από ότι οι υπηρεσίες τις οποίες θέλετε να δημιουργήσετε εσείς στις Βεξέλλες. Λοιπόν, αυτά τα οποία μας είπατε είναι μεν ενδιαφέροντα, μας μιλάτε για συγκεκριμένα αποτελέσματα Κοιτάξτε, ε, ε, αυτά είναι ανακοινώσεις, αυτά είναι σκέψεις, αυτά είναι χαρτιά. Για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε μονόμενα τα στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε, δεν έχετε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά τι αποτρέψαμε, αποτρέψαμε κάτι, γλιτώσαμε από κάτι. Ε, υποτίθεται ότι οι προσπάθειές μας καταπολέμησης ε, των υβριδικών επιθέσεων εμπόδισαν τους ελαικιστές στην Ιταλία, στη Γερμανία ή στη Γαλλία να αναπτύσσονται. Όχι, το αντίθετο συμβαίνει. Συνεπώς λοιπόν αυξήσαμε επίσης την ανθεκτικότητα. Τώρα λέμε για την ανθεκτικότητα στις υβριδικές επιθέσεις. Ε, λοιπόν αυτό δεν αποφασίζεται μέσω μιας γραφειοκρατικής δράσης. Συνεπώς λοιπόν έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για αυτά τα οποία είπατε. Πρώτον γιατί νομίζω ότι υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα νομικού ορισμού. Είναι σαφές ότι όλα τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε, όλες οι συνιστώσεις που δημιουργούν την υβριδική επίθεση είναι τμήματα συμβατικού τύπου επιθέσεων. Επειδή τα συνδυάζουμε όλα τα καθιστούμε υβριδικά. Α, πες ότι το κάνουμε αυτό. Τι κάνουμε, κερδίσαμε κάτι έτσι. Συνεπώς λοιπόν ομολογώ ότι εγώ δεν διακρίνω καμία πρωτοτυπία στην προσπάθειά σας, ε, καμία αποτελεσματικότητα σε ένα θέμα στο οποίο συμφωνώ. Είναι η καλύτερη εναρμόνιση και ο καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι όπως και σε άλλους τομείς η χρησιμότητα των μέσων τα οποία έχετε και θέλετε να δημιουργήσετε είναι η εναρμόνιση εναρμόνιση των βέλτιστων πρακτικών, εναρμόνιση των νομοθεσιών και κατά τα άλλα σας ζητώ συγγνώμη, αλλά κάνουμε τρίχες και δεν έχουμε αποτρέψει πραγματικά τίποτα. Είμαι πάρα πολύ καχύποπτος, ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο ευθύς, αλλά Νομίζω ότι στο Συμβούλιο όλοι τα συζητάνε. Αυτά οι βιδικές επιθέσεις ε, συνεχώς ε, τα έχουμε συζητήσει. Ε, οι βιδικές επιθέσεις επιτρέψτε μου και στον ψυχρό πόλεμο εδώ ήταν. Στην πόλεμο της Ιουκοσλαβίας. Εκεί ήταν. τι έκανε ο Μιλόσεβιτς για πέντε χρόνια. η Υβριδικό πόλεμο έκανε λοιπόν. Τώρα έχουμε πιο περίπλοκα μέσα στη διάθεσή μας αλλά η φύση των εξελίξεων είναι ακριβώς η ίδια και οι προτάσεις τις οποίες κάνετε δεν είναι διόλου μα διόλου πρωτότυπες. Ευχαριστώ τον κύριο Ντονζό και τώρα θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης εδώ μαζί μας. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με το έργο τους και ιδιαίτερα τις εργασίες, ε, το έργο της κυρίας Μογκερίνη, εν περιπτώσει. Ορισμένες φορές έχω την εντύπωση ότι η κυρία Μογκερίνη έχει μια πολιτική απέναντι ε, στην ε, Ρωσική Ομοσπονδία που είναι και μια πηγή των κυβερνόπυλων μια πολιτική λοιπόν αρκετά υποτακτική. Είναι σαν η κυρία Μογκερίνη να μην θέλει, να μην μπορεί ε, να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, φοβάται να περιγράψει αυτές τις απειλές τις ρωσικές, οι οποίες είναι ε, οι πιο πλέον επικίνδυνες. Είναι σαν να μην ξέρουμε ότι ο στόχος της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταρρεύσει. Ένα δισεκατομμύρια ευρώ έλαβε η Stratcom. Είναι, δεν είναι τίποτα για αυτούς. Τίποτα. Ε, δηλαδή το τίμημα είναι αστείο ε, για την υπεράσπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αγαπητοί φίλοι, γιατί ή ακολουθεί αυτή την πολιτική κυρία Μογκερίνη απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολιτική υποτέλεια σε ένα σημείο. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις εκ των προτέρων ε, και τώρα αναμένουμε τις αντιδράσεις σας. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω να μην ξεπεράσετε τα τρία λεπτά ο καθένας θα δώσω το λόγο στην κυρία Κάιν Χούμπερ, όπως προηγουμένως πρώτη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Βεβαίως. Θα απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα για την ενέργεια που τέθηκε. Βεβαίως η ενέργεια, δεν έγινε αναφορά στην ενέργεια, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του, αυτής της, αν την πω, απειλή ε, το Δεν είναι απαραίτητα βέβαια μια δράση η οποία ε, έχει ως σκοπό να αντιστοιχεί σε μια απειλή υβριδικής φύσης όπως τις λέμε εμείς, αλλά υπάρχουν τέτοιες δραστηριότητες, ε, και προφανώς και υπάρχουν ανησυχίε, υπάρχει ο, και άλλο και για την ε, ε, εξασφάλιση του ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο, ε, η προσπάθεια διαφοροποίησης ε, των πηγών ε, ε, ενέργειας. Έχουν γίνει πολλά, όχι πάντα έχοντα κατά νου βέβαια κάποια μορφή υβριδικής απειλής, όμως ε, μιλάμε για μέτρα τα οποία θα μας καταστήσουν πιο ανθεκτικούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιομηχανία της, οι πολίτες της, οι υποδομές της θα είναι πιο ανθεκτικές απέναντι στις απειλές αυτές, είτε τις λέμε υβριδικές ε, είτε όχι. Ε, οπότε, ναι, η απάντηση είναι ναι. Η ασφάλεια των υποδομών σε ό,τι αφορά την ενέργεια, την ενέργεια, τον ανεφοσμό σε ενέργεια, η διαφοροποίηση στις πηγές, ε, είναι σημαντικά στοιχεία, αποτελούν μέρος της κοινή στρατηγικής ε, και του κοινού πλαισίου για την αντιμετώπιση των ευρυδικών απειλών. Και εδώ για άλλη μια φορά υπάρχει θέμα ευαισθητοποίησης για το ποια είναι τα ευάλωτα σημεία, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ετοιμότητα όλων των παραγόντων, ε, όλων των εμπλεκομένων. Αναφέρομαι επίσης στον κανονισμό για την ετοιμότητα απέναντι στον κίνδυνο και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με πληροφορίες, ε, ανταλλαγή πληροφοριών, ε, ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας, ε, όλα αυτά αποτελούν μέρος αυτών των δράσεων. Είναι και η δράση παρθμών 6 του κοινού πλαισίου, νομίζω, το οποίο αναφέρεται μάλιστα ρητά στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριος Μικλόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα για τις υβριδικές απειλές, κατά πόσο υπάρχουν ή όχι, κατά πόσο είναι καλός όρος ή όχι. Ακούστε, υπάρχουν πολλές παρανοήσεις διαρκώς για τις υβριδικές απειλές. Όντως ονομάζουμε τα πάντα υβριδική απειλή, ε, κυβερνοαπειλές κλπ. Καμία δεν είναι υβριδική απειλή από μόνη της μπορεί να αποτελέσουν μέρος μιας υβριδικής εκστρατείας. Ατομικά, μεμονωμένα, η κάθε μία από τις απειλές αυτές δεν είναι υβριδική απειλή, είναι μια μεγάλη διαδήλωση κατά της κυβέρνησης ή μια κυβερνοδραστηριότητα που οδηγεί στο να πέσει ένα, μια ιστοσελίδα της κυβέρνησης ή να δημιουργήσει προβλήματα στο δίκτυο ενέργειας μπορεί να είναι εγκληματικού, ε, εγκληματικής προ, μπορεί να την έχει χρηματοδοτήσει ένα κράτος, από μόνη της όμως δεν είναι ευρυδική. Γίνεται ευρυδική όταν δούμε πίσω από αυτήν και διαπιστώσουμε ότι όλα ε, τα άλλα γεγονότα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης καμπάνιας με, τον ίδιο, με τον ίδιο στόχο. Αυτό τις καθιστά ευρυδικές. Είναι κάτι καινούριο, όχι. Βεβαίω και δεν είναι καινούριο. Αν μιλήσετε στους Ρώσους θα σας πούνε ότι αυτό εμείς το μελετούμε τόσα χρόνια. Ε, με τις ε, ε, χρωματιστές επαναστάσεις ε, στην Ανατολική Ευρώπη. Ε, χρησιμοποιούνται δηλαδή διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί ένα πολιτικό στόχο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που καθιστά σημαντικό να μιλήσουμε για αυτές είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ε, η, ευαισθη, η συνειδητοποίηση από του ε, πολιτικού θύνοντε, από τι διάφορε δομέ μα, ότι πρέπει να μπορούμε να δούμε την ευρύτερη εικόνα, το ευρύτερο πλαίσιο, να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, περιστατικά να δούμε πίσω από αυτά και να δούμε ποια συνοδευτικά μέτρα μπορούν να μα βοηθήσουν να πετύχουμε ποια είναι τα μάλλον τα μέτρα, τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπε δράσεις που έχουν τον ίδιο στόχο. Τώρα για τον ορισμό. Έχουμε νομίζω έναν καλό ορισμό στο κοινό πλαίσιο, σύντομος ορισμός, αλλά αρκετά σαφής για να έχουμε μια κατανόηση του τι μπορεί να συνιστά ευρυδική απειλή. Οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άλλος ορισμός, πιο συγκεκριμένος δηλαδή, μπορεί τελικά να καταστεί αντιπαραγωγικός. Διότι πρόκειται για κάτι το οποίο εξελίσσεται. Εάν εμείς το περιορίσουμε, αν δώσουμε μια συγκεκριμένη, υπερβολικά συγκεκριμένη εικόνα, τότε ξαφνικά μπορεί να βρεθεί εκτό αυτού του πλαισίου ε, μια συγκεκριμένη μορφή δράση. Θα πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε όλα αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεσή μα. Ε, Αυτό λοιπόν είναι καλό για τη συνέχεια, εφόσον το πράξουμε. Τώρα, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις κεντρικοί ε, τομείς που μας δημιουργούν πονοκέφαλο. Ένας είναι η ενέργεια, ο άλλος είναι οι μεταφορές, ο τρίτος είναι η οικονομία, η χρηματοοικονομικός τομέας και ο τρίτος είναι η επικοινωνία. Είναι οι τέσσερις πιο ευάλωτοι τομείς. Ε, ε, και αν δηλαδή εκεί υπάρξει μαζική επίθεση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα για την οικονομία, για την κοινωνία, για την ενέργεια θα θυμάστε πολλοί από εσά, ε, το 2012 είχαμε μια μεγάλη κυβερνοεπίθεση κατά ε, της εταιρείας Ramco όπου 30.000 υπολογιστές ε, σβήστηκαν όλα τα στοιχεία τους και δεν μπορούσε κανείς να τα ανακτήσει. Να ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να μην μας αφήνει να κοιμόμαστε τη νύχτα. Τώρα για το κατά πόσο η υπηρεσία εξωτερική δράση ή ε, ο ύπατο εκπρόσωπο ή το Συμβούλιο είναι αρκετά επικριτικό απέναντι στη Ρωσία, εφόσον η Ρωσία βρίσκεται πίσω από κάποιε από αυτέ τι δραστηριότητε. Εξετάζοντα μια σειρά από μέτρα που έχουν πάρθει, νομίζω ότι έχει καταστεί σαφέ ε, ποιο είναι το συμπέρασμα, ποια είναι η αξιολόγηση που έχει γίνει τη κατάσταση η επιβολή κάποιων κυρώσεων, ε, αντιμέτρων. Ε, είναι πρόβλημα βεβαίως ε, όταν θέλουμε να αποδώσουμε σε κάποιον κάτι. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα όνομα, δηλαδή μια χώρα πίσω από μια τέτοια, μια τέτοια λαβερή δραστηριότητα, εκεί πρέπει να το αποδείξουμε κιόλα. Πρέπει να έχει κανεί στοιχεία αποδεικτικά που να μπορούν να σταθούν και στο δικαστήριο. Είναι δύσκολο η απονομή ευθύνη. Ε, είναι και αυτό μέρο της προσπάθειάς μας βέβαια, έτσι ώστε να καταλάβουν οι πολιτικοί ηθήνοντες ότι σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε δεν υπάρχει απόλυτη και αδιαφυσβήτητη απονομή ε, ευθύνης. Δεν μπορούμε να βρούμε αμέσως το αποδεικτικό στοιχείο, το σαφές. Οι κοινωνίες μας ε, θέλουν οι, κυβερ... οι κυβερνήσεις μας ε, ε, να αναλαμβάνουν συντονισμένη δράση, ακόμα και αν δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποιο είναι ο υπεύθυνο. Και στι κυβερνοεπιθέσει είναι εντελώ αδύνατον αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Πόρτμαν τώρα έχει το λόγο. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποιες από τις ε, απόψεις οι οποίες ακούστηκαν για την παραπληροφόρηση και την αποτελεσματικότητα των απαντήσεων. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις πληροφορίες αυτές είναι πολύ δύσκολο να τους αλλάξει κανείς γνώμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσία ότι είναι προσπάθεια την οποία κάνει για να πείσει η CIA και δεκάδες τέτοιες ιστορίες. Και φυσικά είναι δύσκολο να τους πείσει κανείς να αλλάξουν άποψη. Και δεν προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτό το 10% δεν είναι καν στόχος για μας, αλλά πιστεύουμε ότι το 90% των πολιτών είναι διαθέσιμοι να ακούσουν μια λογική συζήτηση και έχουν ανάγκη η συζήτηση αυτή να ενθαρρυνθεί και μπορούμε να φτάσουμε στους πολίτες αυτούς. Αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο ακολουθούν τα διάφορα κράτη-μέλη, βλέπουμε ποιες είναι οι χρηστές πρακτικές υπήρξαν σαν παράδειγμα, η, παράδειγμα υπόθεση λύσες στην Γερμανία για την υποτιθέμενη απαγωγή μιας μικρής Ρωσίδας από μετανάστες και υπήρξαν δεκάδες χιλιάδες διαμαρτυρόμενοι για ένα έγκλημα που δεν υπήρξε ποτέ. Αντίστοιχα είχε ξεκινήσει μια τέτοια ε, ιστορία στη Λιθουανία που μέσα σε τρεις ώρες αποκαλύφθηκε φυσικά ή αναλήθεια. Είχαν φτιάξει μια ψεύτικη ιστορία για ένα άλλο παιδί που είχε πέσει θύμα απαγωγής από πρόσφυγες. Ε, εδώ είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Δεν κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Υπάρχει ένα όριο σε σχέση με αυτά τα οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε και να πείσουμε ε, μεγάλο ε, κοινό. Ε, μπορούμε, ε, φτάνουμε σε 2 εκατομμύρια πολίτες ε, το μήνα και φυσικά προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και τους ποιοτικού δημοσιογράφους να γράψουν τις δικές τους ιστορίες στη δική τους γλώσσα γιατί μπορούν να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα αν το έχουμε πετύχει αυτό εγώ δεν μπορώ να είμαι απόλυτα αρνητικό Σε σχέση με τα τρία προηγούμενα χρόνια η συζήτηση στην Ευρώπη είναι σαφώς καλύτερη και ποιοτικότερη. Ε, νομίζω ότι έχει υπάρξει υψηλότερη κατανόηση και το επίπεδο της συζήτησης είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Και σε σχέση με τις παρανοήσεις που υπάρχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες ε, ε, μέλη, και στις χώρες εταίρους μπορέσαμε κάποιες παρεμβάσεις να κάνουμε. Σαν παράδειγμα η Γεωργιανή Εκκλησία που είναι ο θεσμός που την χάνει του υψηλότερου σεβασμού στην Γεωργία. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να τους εξηγήσουμε αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Ένωση και αυτό που δεν προσπαθεί να κάνει και είδαμε το ποσοστό των ανθρώπων που δεν εμπιστεύονται την Ένωση να μειώνεται. Συνεπώς λοιπόν οι πόροι πράγματι ε, είναι λίγοι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά πρόοδος έχει υπάρξει. Και για τον πρόεδρο και αυτά τα οποία είπε, να πω ότι η Stratcom είναι η μόνη task force στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει συγκεκριμένη εντολή να ασχολείται με μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και σε σχέση με τους πόρους που έχουμε φέτος είχε γίνει και ε, πέρυσι μια άλλη πρόταση σχετική η οποία δεν ευδοκίμησε να πω ότι είναι ευθύνη όλων να υπάρξει περισσότερο συντονισμός και συνεργασία. Ε, σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν μέρος στη συζήτηση. Πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή ήταν χρήσιμη γιατί θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την παραπληροφόρηση, τα ψεύδη και τις ψευδείς ειδήσει που είναι πολλές φορές πολύ αποτελεσματικά όπλα σε σχέση με άλλα όπλα πραγματικά όπως οι πύραυλοι. Λοιπόν, τελειώνουμε με το 5. Σας ευχαριστώ πολύ. And we can immediately continue to uh, point six of our agenda. Uh, Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τώρα από τους επόμενους ομιλητές να έλθουν εδώ. Έχουμε δύο ομιλητές εκ νέου λοιπόν. σχετικά με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ. summit NATO Λοιπόν, συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε την σημασία που θα έχει αυτή η συνάντηση κορυφής για τη συνέχεια των σχέσεων ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ένωση ο κύριος Σικλόντι και ο κύριος Σελοπτεύσκη. Πρώτα ο κύριος Σικλόντι. Okay, thank you. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, my name is Petra Kolopetsky and I'm... Καλησπέρα σας, Πέτρα Κολοπέτσκι λέγομαι, επικεφαλής ενός τμήματος ε, στην πολιτική διεύθυνση του ΝΑΤΟ, ξέρετε, στο δρόμο για το αεροδρόμιο, στο νέο κτίριο. Έχουμε μετακομίσει εκεί εδώ και κάποιες εβδομάδες, πάρα πολύ ωραίο. Και έχουμε τη σύνοδο σε κανένα μήνα και θα σας ενημερώσω σύντομα για το τι θα συζητηθεί σε αυτήν την σύνοδο 11 και 12 Ιουλίου. Θα έχουμε βασικά θέματα που θα συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Πρώτα απ' όλα άμυνα και αποτροπή. Η άμυνα και η αποτροπή είναι προφανώς ο σκοπός του ΝΑΤΟ από το 1949 και ακριβώς ε, το θέμα αφορά τους συμμάχους ε, και τους φίλους ε, στη συγκεκριμένη περίοδο το θέμα ακριβώς αφορά την προκεχωρημένη παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη κάτι θα έχετε ακούσει αποτέλεσμα δράσεων του ΝΑΤΟ από το 2014 και 2015 και εδώ ως αντίδραση στην επιθετικότητα της Ρωσίας στην Κρυμαία, στην Ουκρανία. Μάλλον θα έχετε ακούσει ότι το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αναπτύξει κάποιες ε, συμβολικές ε, δυνάμεις, μονάδες ε, απολύτως αναλογικές στο ανατολικό κομμάτι της επικράτειας των συμμάχων, στις βαλτικές δημοκρατίες δηλαδή, Βουλγαρία, Πολωνία και Ουγγαρία και Σλοβακία. Λοιπόν, αυτό ακριβώς θέλουμε να δούμε φέτος και τα επόμενα έτη, να δούμε δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε αυτές τις ε, μονάδες που μέχρι στιγμής είναι συμβολικές εάν αυτό απαιτηθεί για να υπερασπιστούμε ή για να αποτρέψουμε μια επίθεση. Αυτά θα συζητήσουμε στο κομμάτι άμυνας και αποτροπής. Το ένα είναι αυτό. Δεύτερο, που θα συζητήσουν οι ηγέτες είναι κάτι το οποίο λέμε προβολή σταθερότητας εμείς στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή προσπαθούμε να προβάλλουμε κάποιο επίπεδο σταθερότητας στην γειτονιά μας, κυρίως προς Ανατολάς και προς Νότον, με διάφορα μέσα, αλλά κυρίως την εκπαίδευση και αυτό το οποίο λέμε βεβαίως ενίσχυση των εταίρων μας, όχι οπωσδήποτε μελών μας, όπως η Ουκρανία, η Γεωργία, η Μολδαβία, αλλά και η Ορδανία, η Τινησία στο Νότο, ίσως και η Λιβύη ακόμα στο μέλλον, για να μπορέσουν να υπερασπίσουν αυτούς απέναντι σε διάφορες απειλές και υβριδικές απειλές επί τη ευκαιρία μόνες τους να μην χρειάζεται δηλαδή το ΝΑΤΟ να αναπτύσσει στρατεύματα και πόρους για να σταθεροποιηθούν αυτές οι περιοχές στην γειτονιά μας. Αυτό είναι το πακέτο προβολής σταθερότητας, όπως λέμε, και θα δείτε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα στο θέμα αυτό, ε, υπό μορφή ε, ενισχυμένης, ε, θα έλεγα, συνεργασίας με την Ιορδανία, ενός πακέτου αρχικού με την Τινησία και ενισχυμένης εκπαίδευσης ε, και στο Ιράκ που πιθανότατα θα ανακοινώσουμε τον Ιούλιο. Αυτό θα είναι το υπαριθμόν 2, το υπαριθμόν 3 το θέμα είναι οι σχέσεις με την Ένωση και νομίζω ότι θα επεκταθούμε σε αυτό. Ξέρετε τώρα έχουμε 74 συγκεκριμένους τομείς ε, που έχουμε ανοιχνεύσει ως ε, τομείς συνεργασίας, τομείς οι οποίοι καλύπτουν μια σειρά θεμάτων ε, υβριδικά κυβερνοάμυνα, οικοδόμηση δυνατοτήτων αλλά και ζητήματα στρατιωτικής κινητικότητας που ήδη έχετε αναφέρει. Αντιτρομοκρατία κτλ. Ε, πολλά πράγματα λοιπόν και αυτή τη στιγμή 22 μέλη, κράτη είναι μέλη και των δύο οργανισμών. Ε, εντάξει, δεν είναι όλα τέλεια. Ρίχασαμε πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και δύο χρόνια. Και βεβαίως ένα υποθέμα αυτών των φακέλων θα είναι ο υβριδικός ε, πόλεμος. Μιλήσατε λίγο για το τι εστί υβριδικός πόλεμος, αν είναι νέα ή παλιό, αν πρέπει να το λέμε υβριδικό ή όχι. Και βεβαίως ε, η υβριδικότητα του πράγματος είναι ακριβώς ο συνδυασμός των απειλών και από καιρού εις καιρών, όπως είδατε και στην Ουκρανία, έχουμε ακριβώς ε, στον ορίζοντα αυτήν την μεγάλη στρατιωτική δύναμη που δίνει ακριβώς μια διαφορετική χρειά και στις μη στρατιωτικές ε, δράσεις ε, θα έλεγα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τέταρτο θέμα οπωσδήποτε είναι αυτό το οποίο λέμε εξυγχρονισμός του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ πάντα ξέρετε ότι προσαρμόζεται. Μέχρι το 1990 στόχος ήταν συλλογική άμυνα, μετά πέρασε σε θέματα στάθεια στην γειτονιά μας, ε, Βαλκανική πόλεμη, μετά είχαμε την αντιτρομοκρατία, επιχειρήσεις εκτός περιοχής ευθύνης και παρερχόμαστε τώρα στην συλλογική άμυνα με την επιθετικότητα της Ρωσίας κάποια έτσι παραδοσιακά θα έλεγα ζητήματα με παραδοσιακά στρατιωτικά μέσα. Το ΝΑΤΟ λοιπόν συνεχώς ε, προσαρμόζεται για να είναι πιο αποτελεσματικό, για να λαμβάνει αποφάσεις πιο γρήγορα με τρόπο αποτελεσματικό. Αυτό θα είναι το κομμάτι του εξυγχρονισμού και ένα κομμάτι βεβαίως είναι ακριβώς η προσαρμογή της δομής ε, διοίκησης. Θα έχετε ακούσει ότι έχουμε κάποιες νέες διοίκησεις. Ε, μία φορά τον Βόρειο Ατλαντικό, η άλλη είναι η διοίκηση της επιμελητίας ε, που θα βασίζεται στη Γερμανία. Και τέλος θα μιλάσουμε και για τον διαμοιρασμό του βάρους. Θα έχετε ακούσει τον πρόεδρο Τραμπ που παραπονιέται ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ξοδεύουν και πολλά στην άμυνα. Ξέρετε ότι υπάρχει μια κατευθυντήρια γραμμή για 2% του ΑΕΠ. Δεν υπάρχουν πολλές χώρες που φτάνουν στο 2%. Γύρω στις 7 φέτος ε, ήταν πριν από δύο χρόνια ήταν μόλις 3. Οπότε νομίζω ότι αλλάζουν τα πράγματα. Προφανώς γνωρίζετε ότι υπάρχει κάτι το οποίο λέμε δέσμευση δαπανών για την άμυνα δηλαδή κάθε σύμμαχος θα προσπαθήσει να φτάσει το 2% μέχρι το 2025 μπορώ να σας πω ευθύς αμέσως ότι δεν θα το καταφέρουν αυτό όλοι μόλις ακούσαμε την κυρία Μέρκελ την ε, προηγούμενη εβδομάδα που είπε ότι η Γερμανία θα είναι στο 1,5% το 2025 το οποίο σε απόλυτους αριθμούς βεβαίως δεδομένου του γερμανικού ΑΕΠ είναι ένα τεράστιο νούμερο, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι 2%. Και νομίζουμε ότι οι Αμερικανοί φίλοι μας θα μας πούν τον Ιούλιο ότι αναμένουν κάποια περισσότερα. Αυτό λοιπόν θα είναι το πέμπτο θέμα. Είμαι σίγουρος ότι κάποια αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα του αποδώσουν μεγάλη σημασία. Οπότε θα σταματήσω εδώ. Όπως είδατε από αυτά τα θέματα βλέπετε ότι αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώ αναμένουμε την περαιτέρω συνεργασία στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο τώρα στον επόμενο μιλητή θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εδώ και τρία χρόνια όταν ε, είχαμε συμφωνήσει ε, για τη σχέση με τον ΝΑΤΟ, μας είχαν κατηγορήσει ότι είχαμε μια κάποια μορφή ζήλιας απέναντι στο ΝΑΤΟ ή επειδή θέλαμε να δημιουργήσουμε μια δική μας, ένα δικό μας σύστημα στον τομέα της άμυνας. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια κοινή πλατφόρμα και να υπάρξει μια πραγματική συνεργασία ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη μορφή αυτής συνεργασίας κύριε Τελουπέτσκι, αναφερθήκατε επίσης ε, και σε μια ομάδα χωρών όπως οι Βαλτικές χώρες και η Πολωνία που συνεργάζονται πλέον στενά, είναι ένα νέο βήμα προς τα εμπρός ε, και είναι μια νέα μορφή αλληλεγγύης ε, από τις χώρες που απειλούνται από τη Ρωσία και μάλιστα με υβριδικό τρόπο. Ο επόμενος ομιλητής, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνάντηση του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο είναι μια συνάντηση του ΝΑΤΟ και είναι σωστό το, το κύριο Τσελουμέσκι τα παρουσίασε σωστά. Να προσπαθήσουμε να δούμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, να δούμε τι περιμένουμε. Καταρχάς ένα γενικό σχόλιο. Αν το ΝΑΤΟ πραγματικά είναι ικανό, ισχυρό, ευέλικτο ε, να διασφαλίσει τις ε, υποχρεώσεις στον τομέα της συλλογικής άμυνας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα καταστήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ισχυρή. 22 χώρες μέλη είναι ε, φυσικά και μέλη του ΝΑΤΟ και αυτό και μέσα είναι στην συνθήκη ότι οι 22 αυτές χώρες τουλάχιστον θα ήθελαν να δούνε την ασφάλειά τους να γίνεται αντικείμενο εγγύησης από την ίδια τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Πέραν όμως αυτών των 22, ένα ισχυρό ΝΑΤΟ είναι προς το συμφέρον όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Τώρα τι περιμένουμε εμείς ε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπατε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει την πορεία να εντείνει τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, έχει γίνει θέμα προτεραιότητας και υπάρχουν σοβαρές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν αναλυφθεί, που έχουν ξεκινήσει πλέον να εφαρμόζονται όπως και η μόνιμη διαδρομένη συνεργασία στον στρατιωτικό ταμέα και οι πρωτοβουλίες τύπου LEAD. Τώρα το αν μαζιλεύει ή όχι το ΝΑΤΟ αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Να μην ξεχνάμε ότι μέσα από τις προσπάθειες αυτές και την ανάπτυξη των στρατιωτικών ικανοτήτων και με την ανάπτυξη της ε, λειτουργικής διαθεσιμότητας των στρατιωτικών μέσων. Οι, τα μέσα αυτά δεν νοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στις χώρες μέλη. Ως εκ τούτου όλες αυτές οι δυνατότητες οι στρατοτικές δημιουργήθηκαν με την βοήθεια και συνεργασία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ε, καθίστανται διαθέσιμα ανάλογα με τις πολιτικές επιθυμίες και αποφάσεις ε, της Ένωσης και του ΝΑΤΟ που θα γίνονται αποδεκτές σε εθνικό επίπεδο. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα το οποίο θα θέλαμε εμείς να βγει ε, εκ των προτέρων θα έλεγα στη συνάντηση αυτή κορυφής του ΝΑΤΟ. Στηρίζουμε λοιπόν τις αυξημένες δυνατότητες της ευρωπαϊκής πλευράς έτσι ώστε να δημιουργήσει επιπλέον τέτοιες δυνατότητες και να αυξήσει τις λειτουργικές ικανότητες των στρατιωτικών μας δυνάμεων. Τέτοιου είδους αναγνώριση θα βοηθήσει φυσικά και το ΝΑΤΟ έμεσα, δηλαδή αν αυξήσει κανείς τις εθνικές δυνατότητες αυξάνονται ε, και οι δυνατότητες να ωφεληθεί το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ανακοινωθέν της συνάντησης κορυφής. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα. Και έρχομαι εδώ τώρα στο δεύτερο σημείο, το, το μήνυμα ενότητας που πρέπει να στείλουμε. Ένα τέτοιο μήνυμα είναι ένα μήνυμα ενότητας σε σχέση με τους στόχους. Είναι κάτι το σημαντικό και για το ίδιο το κοινό μας που πρέπει να καταλάβει ότι το μέσο αυτό, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, συνεργάζονται έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρα στους στόχους που επιθυμούν, καλύτερη άμυνα, καλύτερη διαχειριστική ικανότητα των κρίσεων και αντίδρασης στις απειλές οι οποίες ε, έρχονται στην επιφάνεια. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το κοινό το δικό μας, αλλά και τους πιθανούς ε, αντιπάλους, είτε τους ονοματίσουμε είτε όχι. Πάντως, ε, είναι θα έλεγα πολιτικές οι οποίες είναι απαραίτητες και έχουμε μπροστά μας ε, ε, τα μέσα τα οποία συνολικά διατίθενται είτε σε επίπεδο διπλωματικό είτε σε επίπεδο στρατιωτικό, δηλαδή είτε κυρώσεις είτε επιμέρους άλλες στρατιωτικές δράσεις. Το βασικό και στις δύο περιπτώσεις είναι η ενότητα. Και η τρίτη παρατήρηση αφορά στο μέλλον. Έχουν υπάρξει 74 προτάσεις σε μια σχετικά σύντομη χρονική περίοδο, διετή χρονική περίοδο. Καλό θα είναι ίσως ε, να μείνουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις προτάσεις οι οποίες ε, πράγματι θα είναι ε, χρήσιμες. Μία επιπλέον προσδοκία από τη συνάντηση κορυφής λοιπόν είναι να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε πρακτικά συγκεκριμένα μέσα τα οποία θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε συντονισμένες μορφές απάντησης και ανταπόκρισης. Θέλουμε συγκεκριμένες δράσεις. Να πω κάποιους από τους τομείς τους οποίους είτε βραχυπρόθεσμα είτε μεσοπρόθεσμα μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Καταρχάς, στρατιωτική κινητικότητα. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα και για τις δύο πλευρές. Να μπορέσει, για να μπορέσει το ΝΑΤΟ να καλύψει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να λειτουργήσει στρατιωτικά, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα μετακίνησης των στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό δεν τον επιθυμεί η Ένωση, δεν το επιθυμεί το ΝΑΤΟ. Τα κράτη-μέλη το επιθυμών Θέλουν στην περίπτωση που υποστούν επιθέσεις να τύχουν συνδρομή στρατιωτικής γρήγορα. Και επίσης αν θέλουν να ξεκινήσουν μια δράση μακράν της Ένωσης θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα για να το κάνουν αυτό. Συνεπώς νομίζω ότι η στρατιωτική κινητικότητα είναι η βασική αν θέλετε προτεραιότητά μας. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της διαλειτουργικότητας. Να σας ε, αναφέρω δύο περιπτώσεις παραδείγματα. Η Βοσνία, σαν παράδειγμα, ε, το, Βερολίνο ΣΥΝ δηλαδή, διαδικασία Βερολίνο ΣΥΝ, ε, υπό την διοίκηση του ε, αντιστράτηγου του στρατηγίου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Έχουν λοιπόν εδώ εντοπιστεί συγκεκριμένοι τομείς στους οποίους ε, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εμπλοκής ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν παράδειγμα η επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση μάλλον Έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση 170 τέτοιες περιπτώσεις. Το ΝΑΤΟ θα το έκανε καλύτερα βρήκαμε εκ των υστέρων γιατί ε, ήταν υπεύθυνη για τη στρατηγική η οποία ακολουθείται σε, στην Βοσνία. Θα πρέπει λοιπόν οι στόχοι να επιδιώκονται με τα σωστότερα δυνατά μέσα. Μετά από κάποια χρόνια στη Βοσνία φάνηκε ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή δράση στα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία είναι υψηλής προτεραιότητας και τώρα πάλι και θέλουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε ασφάλεια στην περιοχή έτσι ώστε οι χώρες της περιοχής να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες απαιτείται να γίνουν. Δεύτερη περίπτωση, το Ιράκ. Το Ιράκ θα αναπτύξει, μάλλον το ΝΑΤΟ θα αναπτύξει μια συμβουλευτική ομάδα στο Ιράκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναπτύξει μια διερευνητική ομάδα και ε, συνεχίζει η εντολή της μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Ε, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε, να μπορέσουμε δηλαδή να συντονίσουμε και την υπάρχουσα φάση προγραμματισμού και όχι να περιμένουμε να πάνε και οι δύο αποστολές εκεί και εκ των υστέρων να τις συντονίσουμε. Είναι μια καλή θα έλεγα ευκαιρία να βγάλουμε συμπεράσματα για το μέλλον. Φυσικά οι υβριδικές επιθέσεις είναι προτεραιότητέ μας, είναι θα έλεγα τα τελευταία τέσσερα χρόνια προτεραιότητα του ΝΑΤΟ και θα παραμείνει κάτι τέτοιο και στο μέλλον. Μόνο μέσω της σωστής αλληλοεπίδρασης οι χώρες μας θα μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Μια τρίτη προσπάθεια, το είχα πει και πέρυσι, είχαμε μια δράση του ΝΑΤΟ και ε, με μια συμπληρωματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος είναι ακριβώς το αντίθετο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε γυμνάσια, να προσπαθούμε να εντοπίζουμε ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι οι επικαλύψεις και να προσπαθήσουμε να ανασχεδιάσουμε ε, τους μηχανισμούς ανταπόκρισής μας αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές σειράξεις τις οποίες θα μπορούσε να παρέμβει το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνουν σε ένα πλαίσιο υβριδικό. Και τέλος η εταιρική αν θέλετε βελτίωση των ικανοτήτων. Αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ κάποιος ο Πίτερ, το DCBI και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί και ε, να βοηθήσει στον τομέα αυτό τις γειτονικέ χώρες. Ήδη υπάρχουν γεωγραφικά εντοπισμένες περιοχές. Μπορούμε εκεί να κάνουμε ε, διάφορα βήματα συνεργασίας. Μολδαβία, Γεωργία, Ουκρανία είναι ο ένας χώρος. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ο δεύτερος χώρος και εκεί πρέπει να τους βοηθήσουμε και τρίτον κάποιες χώρες του Νότου αναφερθήκατε στην Ιορδανία και είναι για μας βασική προτεραιότητα σε ορισμένες χώρες, σε ορισμένα θέατρα είναι σημαντικό να πάμε εκεί συνεργαζόμενοι και με κοινή σημαία. Σε κάποιες άλλες χώρες κάτι τέτοιο δεν θα ήταν παραγωγικό. Εκεί θα ήταν καλύτερα να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε με πιο διακριτικό τρόπο να λειτουργήσουμε. Ένα ακόμα πράγμα, η πρόοδος ε, που απαιτείται να γίνει σε κάποιους τομείς και ε, υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Μετά έχουμε το θέμα της ε, καταπολέμησης του, της τρομοκρατίας. Εδώ θα πρέπει να εντοπίσουμε ακόμα το τι μπορούν να κάνουν μεμονωμένα και συλλογικά οι δύο οργανώσεις. Δεν είναι εύκολο, δεν ιδιαίτερα για το ΝΑΤΟ είναι δύσκολο και τέλος να προσπαθήσουμε να δούμε αν σε ορισμένους τομείς, σε ορισμένους χώρους ε, θα ήταν ε, λογικό να υπάρχουν κοινέ δυνάμεις σε σχέση με την παροχή και διασφάλιση ειρήνης και ασφάλειας νομίζω ότι και στα πλαίσια των προτεραιοτήτων τις οποίες έχουμε ορίσει και στα πλαίσια της συνεργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη οι βασικές αρχές ισχύουν. Το θέμα είναι πώς θα τις καταστήσουμε λειτουργικές. Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε πρακτικά βήματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν παράδειγμα μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε εμεί σε όλες τις αποστολές δώσει συμβούλους για θέματα φύλου. Και νομίζω ότι πώς μπορούμε να τα καταστήσουμε αυτά πιο λειτουργικά. Uh, uh, Πολύ δουλειά επίσης με ΜΚΟ. Είναι μια πηγή έμπνευση για μας, διότι ότι συχνά αυτοί βρίσκονται εκεί, επιτόπου, συλλέγουν τις πληροφορίες για το τι χρειάζεται. Θα σταματήσω κάπου εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κλόντι. Αναφερθήκατε στο θέμα της ορατότητας και είπατε ότι υπάρχει θέμα ορατότητας των στρατιωτικών δυνάμεων. Αναφερθήκατε και στις διάφορες απειλές. Εκ μέρους της Ρωσικής Μοσπονδίας, παραδείγματος χάρη. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι οι πολιτικοί εκπρόσωποι της Ρωσίας, αλλά και οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει επίδειξη δύναμης. ο πρόεδρος Ρίγκαν είναι αυτός ο οποίος κέρδισε τον ψυχρό πόλεμα, πόλεμο. Και παρόλα αυτά χαίρει μεγάλης εκτίμησης στη Ρωσία και έχει τιμηθεί εκεί. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση λοιπόν. Πρέπει να μπορούμε να επιδεικνύουμε την ισχύ μας, να την δείχνουμε. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για πρόσφατες, ε, πρόσφατα γεγονότα όπως αυτά της Ουκρανίας. Κύριε Γιούρεκ, θέλετε να θέσετε κάποιο ερώτημα, θέλετε να σχολιάσετε. Ναι, ευχαριστώ. Άκουσα μόνο το τέλος, ε, διότι ε, η πτήση μου άρχισε δυόμιση ώρες. Οπότε ελπίζω να μην θέσω ερωτήματα που έχουν ήδη απαντηθεί. Ήθελα να ρωτήσω αντιδράσω λοιπόν σε αυτά που ακούστηκαν, αλλά θέλω να πω κάτι για τον Nord Stream 2. Έγινε αναφορά στο Nord Stream 2. Όχι. Ωραία. Ε, κανένα άλλο θέμα δεν είναι τόσο κοντά, δεν αφορά τόσο πολύ τη σχέση μεταξύ της άμυνας ε, και της αλληλεγγύης, αλλά και το πολιτικό σκέλος. Ε, διότι αν δεν μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, εάν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή κάνουν μια ενεργειακή εισβολή και διχάζουν την Ευρώπη, χωρίζουν την Ευρώπη στα δύο. Υπάρχει ήδη μια απομόνωση με τον Nord Stream 1 και τώρα θα υπάρξει μια δεύτερη απομόνωση με τον Nord Stream 2. Εάν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό, αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητε άμυνά μα είναι πολύ ισχνές. Αναφέρομαι τώρα στην Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ αφορά ε, το στρατιωτικό σκέλος, βεβαίως. Ένα άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι είχαμε, έχουμε και το ζήτημα της συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που έχει διακοπεί και πολλές εταιρείε σκέφτονται κατά πόσο πρέπει να ανοίξουν παρεδόση με το Ιράν. Φοβούνται τις αντιδράσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης ε, δεν δείχνει αυτό ουσιαστικά με δραματικό τρόπο το πόσο αδύναμη είναι η πολιτική μας. Αν φοβούνται ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επιχειρήσουν με το Ιράν λόγω μιας μονομερούς απόφασης των Αμερικανών, του Αμερικανού Προέδρου. Και ξεχνάμε ξαφνικά την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη παρά τις τόσες δηλώσεις ε, των Ευρωπαίων ηγετών. Θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για αυτά τα δύο ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιούρεκ. Λοιπόν, ποιος ε, θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ναι. Ε, ε, ε Κοιτάξτε, είναι εύκολη απάντηση θα έλεγα γιατί δεν μας απασχολεί τόσο πολύ ο Nord Stream 2 και το Ιράν στο το αλλά να κάνω κάποια σχόλια. Έχετε απόλυτο δίκιο είναι θα έλεγα μια σφίνα στόχο έχει να διχάσει τους Ευρωπαίους συμμάχους εδώ κάποια κράτη-μέλη της Ένωσης από πλευράς Ρωσίας όπως και ο 1 ήταν κάποια στιγμή ταυτόχρονα νομίζω ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες να σταματήσουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Υπάρχουν πολλά χρήματα στην υπόθεση αυτή και βούληση από διάφορες πλευρές και ξέρω αν υπάρχει τρόπος να υπερβούμε αυτή την απομόνωση που υπάρχει δηλαδή να απομονώσουμε την κεντρική και ανατολική Ευρώπη από τις πιο επικέρδεις ε, δυτικοευρωπαϊκές αγορές γιατί το αέριο Ξέρετε, δεν έχει ενιαία τιμή, διαφέρει από αγορά σε αγορά. Και αυτό ακριβώς είναι και το θέμα. Μία λύση είναι οι εναλλακτικέ ε, πηγές ε, και διοδι μεταφορών ε, και προμηθευτές όσα περισσότερα τέρμινα λιγροποιημένο φυσικό αερίο έχουμε τόσο το καλύτερο όσο περισσότερο αμερικανικό αέριο έρχεται στην Ευρώπη τόσο το καλύτερο όσο μεγαλύτερος ανταγωνισμός ε, υπάρχει τόσο το καλύτερο και νομίζω πως η ε, Ρωσία αισθάνεται την πίεση των Αμερικανών ε, των διαφόρων τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου με την έννοια ότι μειώνονται οι τιμές, αλλάζουν οι διαπραγματευτικές τακτικές. Αν και το ΝΑΤΟ προφανώς παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγορές ενέργειας, δεν είναι κάτι το οποίο ε, μας απασχολεί ε, συγκεκριμένα. Όσον αφορά τα ζητήματα του Ιράν, ε, πράγματι τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά γιατί ασχολούμαστε με προσπάθειες μη διάδοσης ε, των πυρηνικών σε ολόκληρη την εφήλιο και παρακολουθούμε στενά ακριβώ και τη σχετική συνθήκη, τα πυρηνικά προγράμματα και τους περιορισμούς τους, τα πυραυλικά προγράμματα. Η κατάσταση τώρα δεν είναι ιδιώδης. Ε, ότι πιθανώ το ατυχέστερο κομμάτι είναι ότι αν αποσυρθούν όντω οι ευρωπαϊκές εταιρείε από εκεί, κάποιε άλλες εταιρείε θα γεμίσουν το κενό, οι ρωσικέ εταιρείε και οι κινέζικες. Και αυτό νομίζω είναι το χειρότερο δυνατό σενάριο. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια επαναδιαπραγμάτευση τουλάχιστον μεταξύ των δυτικών μερών της ε, συμφωνίας ε, για να βρεθεί μια λύση αλλά όπως είπατε είναι μια τυχής ε, κατάσταση και το ΝΑΤΟ πέρα από το να παρακολουθεί τις εξελίξεις δεν έχει εμπλακεί τόσο πολύ στο θέμα αυτά μπορώ να πω από αυτό νομίζω ότι λίγα έχουμε να προσθέσουμε σε αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος για την ενεργειακή ασφάλεια βεβαίως υπάρχουν σοβαρές ε, συνέπειες ε, που αφορούν την ασφάλεια ε, πραγματικά το καλύτερο μέσο είναι μια διαφοροποίηση των πηγών και σας το είπα, σας το ανέφερα και πριν υπάρχει ακριβώς ένας έλεγχος που κάνουμε και εξετάζουμε τις διάφορες ευπάθειες. Αν υπάρχει μια εξάρτηση κατά 100% από μία πηγή, αυτό από μόνο του είναι ένα σημείο αδυναμίας. Βεβαίω ε, οι εναλλακτικές ε, πηγές ε, και διαδρομή είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και ε, βεβαίω μπορούμε να έχουμε μία σχέση που ε, εντάξει μπορεί να είναι με κάποιον ε, πολιτικό ανταγωνιστή στο πολιτικό επίπεδο αλλά μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος στον τομέα της ενέργειας δηλαδή το ένα δεν σημαίνει απαραίτητα και το άλλο Παρ' όλα αυτά η διαφοροποίηση των πηγών έχει μεγάλη σημασία εκεί πέρα Συμφωνώ πλήρω. Και βεβαίω είναι μια συζήτηση η οποία θα συνεχιστεί για καιρό θα ε, γίνει ή θα γίνουν τέτοιες συμφωνίες ε, και στο μέλλον και μπορούμε μόνο να προσπαθήσουμε να έρθουμε ως το δυνατόν πιο κοντά σε μια ιδεώδη κατάσταση και οπωσδήποτε και η ασφάλεια έχει μεγάλη σημασία. Βεβαίω, έχει μεγάλη σημασία για κάποιες χώρες, κάποιες προσεγγίσεις, ίσως λιγότερο για άλλες. Και βεβαίω ε, κάποια συμφέροντα θα έλεγα θα πρέπει να τεθούν στο προσκήνιο. Για το Ιράν λίγα έχω να προσθέσω. Και βεβαίω ε, υπάρχει ακριβώ αυτή η δυσαρέσκεια για το ότι οι ΙΠΑ επέλεξαν να μην ε, σεβαστούν τη συμφωνία. Είναι κάτι το οποίο πράγματι έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια ειδικά μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιριών θυμάμαι, άκουσα κάτι νούμερα της τάξης των 14 έως 20 δισεκατομμυρίων και αύξηση του εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Μια πολύ ευαίσθητη εξέλιξη. Το αμερικανικό εμπορίο είναι γύρω στα 600 εκατομμύρια, αν άκουσα καλά. Οπότε προφανώς ε, θα βλάψει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και κάποιες εταιρείε θα πρέπει να κάνουν μια επιλογή. είτε θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με το Ιράν είτε με την Αμερικανική αγορά. Δύσκολες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν. Οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν λίγο, αλλά ουσιαστικά το πρόβλημα υπάρχει. Και βεβαίως το θέμα είναι ποιος θα αναπληρώσει αυτό το κενό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλατε να πείτε κάτι. Δυστυχώς ε, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει χρόνος ε, για περαιτέρω συζήτηση. Ε, έχετε ένα λεπτό, Πλέον ο πρόεδρος, οι διερμηνείς τελειώνουν σε ένα λεπτό. Οι διερμηνείς όμως τελειώνουν σε μισή ώρα το ωράριό μας. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω, απευθύνομαι στον κύριο Κλούτη γενικός κανόνας είναι ότι οι πολιτικοί ανταγωνιστές ε, βεβαίω μπορεί να είναι ε, αξιόπιστοι εταίροι στην ενέργεια. Μα δεν είναι ανταγωνιστή. η Ρωσία, παραβιάζει ε, τους διεθνείς κανόνες και έχει βάλει στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας. Ε, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία να ακούσουμε τις εξηγήσεις αυτές. Ευχαριστώ την ε, Γραμματεία και τους διερμηνείς. Η Επιτροπή μας ε, θα συνεχίσει τη συνεδρίαση αύριο, 9.30. Ναι, αλλά εγώ θέλω μια απάντηση. να, απαντήσετε στον, κύριο, να απαντήσει στον κύριο Γιούρεκ. Ναι, βεβαίω. Και μετά τη συνάντηση μπορούμε να το πούμε και διμερώς. Ε, ανταγωνιστής, ε, πολιτικός ανταγωνιστής δηλαδή, ε, στην περιοχή, στη γειτονιά μα, ναι βεβαίω, πολιτικό ανταγωνιστή. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή και γι' αυτό ίσως να πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο. Και ποια είναι η εναλλακτική σα τελικά, η δική εναλλακτική τι είναι, να απομονώσουμε τη χώρα αυτή τελείως διότι έχει κάνει κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν και έχει παραβιάσει θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής ασφάλειας και ως, ε, ε, και ως ε, απάντηση τι πρέπει να κάνουμε εμείς, να κόψουμε οποιοδήποτε, οποιοδήποτε δεσμό αυτή τη χώρα δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να σας απαντήσω εγώ σε 30 δευτερόλεπτα στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ τον κύριο Γιούρεξ, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Είχαμε πει 6, πήγαμε λίγο παραπέρα. Θα τα πούμε αύριο στις 9.30. Καλό βράδυ.